Καθίστε παρακαλώ για να ξεκινήσουμε για σήμερα. Καλή σας ημέρα λοιπόν, να καλωσορίσω όλους ιδιαίτερους ε, τους προσκεκλημένους μας, οι οποίοι θα λάβουν και το λόγο στη μικρή ακρόαση που έχουμε σήμερα για την παράνομη αλία. Σημείο 9 της ημερήσιας διάταξη έκθεση Λέβιν κατά πολέμηση της παράνομης αλίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Όπως γνωρίζετε, έγινε ήδη ανταλλαγή απόψεων τον Οκτώβριο. 26 Ιανουαρίου η κυρία Λέβιν παρουσίασε το προσχέδιο του εγγράφου εργασία τη και τον Απρίλιο επίση μα παρουσίασε το δεύτερο εγγράφο εργασία τη κυρία Λέβεν. Σήμερα μετά την ε, υπόδειξη και το αίτημα της εισηγήτριας ε, θα έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων με εξέχοντες εκπροσώπους από τις ΙΠΑ και από την Ιαπωνία. Επιρρογνώμες μεταξύ άλλων ε, για την παράνομη αλία Επειδή ήμουν στην ε, Παγκόσμια Οργάνωση Αλίας Σάικα γνωρίζω προσωπικά τους ε, αξιότιμους ε, προσκεκλημένους μας. Θέλω να σας καλωσορίσω όλους ιδιαίτερως. Είστε δύο αντιπροσωπείες που πάντοτε έχετε διακριθεί για την, τον αγώνα που δίνετε κατά της παράνομης αλίας. Θα δώσω όμως καταρχάς το λόγο στην εισηγήτρια για να ξεκινήσουμε έτσι τη συζήτηση και μετά θα δώσω το λόγο στις δύο αντιπροσωπείες. 15 λεπτά θα έχουν στη διάθεσή τους και θα ακολουθήσει ανταλλαγή απόψεων με όλους τους βουλευτές της Επιτροπής μου. Κυρία Λέβιν, έχετε το λόγο. Thank you very much, Madam Chair. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι που μπορούμε για μια ακόμη φορά να συζητήσουμε την έκθεση αυτή Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδες εισηγητές, με τους οποίους είχα διμερείς συναντήσεις, με τους περισσότερους από αυτούς. Και συζητήσαμε κάποιες από τις τροπολογίες. Για να μπορέσουμε όμως αυτή τη φορά να συζητήσουμε παρουσία δύο εξεχόντων ε, εκπροσώπων δύο άλλων ε, σημαντικών παγκόσμιων ε, αλληλευτικών αγορών και με τη δόκτωρα Ρεμπέκα Λέντς που είναι διευθύντρια του Γραφείου των Εθνών Υποθέσεων του ΝΟΑ, οργανισμού ε, από τις είπα και με τον κύριο Μασανόρη Μιαχάρα που είναι ο ε, Διευθύνος Σύμβουλος του Αλληλευτικού Οργανισμού της Ιαπωνίας για να ε, μπορέσουμε λοιπόν να συζητήσουμε και έχουμε καλέσει βέβαια και εκπρόσωπο από την Κίνα μια ακόμη παγκόσμια υπερδύναμη που είναι και χώρα που παράγει τα περισσότερα αλληλευτικά προϊόντα. Επί του παρόντος βέβαια δεν ε, καταφέραμε να έχουμε θετική απάντηση από την, ε, από την Κίνα, ούτε ε, υπήρχε δυνατότητα βιντεοδιάσκεψης ή να έρθει κάποιος εδώ στις Βρυξέλλες. Δεν μπορούσε να στείλει κανέναν και η αντιπροσωπεία της Κίνας στις Βρυξέλλες. Και πραγματικά με λυπεί αυτό, γιατί αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε την παράνομη έλλειψη σε παγκόσμιο επίπεδο, μπορούμε αυτό να το πετύχουμε μόνο αν συνενωθούν και συσπηρώσουν τι προσπάθειέ του όλοι οι παγκόσμιοι εταίροι. Για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να καταπολεμήσουμε αυτό το παγκόσμιο φαινόμενο, αυτή την παγκόσμια μάστιγα. Κυρία Λέντ και κύριος Μιαχάρα όμως έχουν διαβάσει την έκθεσή μου και πραγματικά περιμένω με ανυπομονησία να ακούσω τις ε, δικές τους απόψεις σε σχέση με τις προτάσεις μας. Παραδείγματο χάρη, πρόταση περί υποχρεωτικής ανεξάρτητης ανεξάρτητης τακτικής αξιολόγησης ή επέκταση της εντολής ε, των RFMOs ε, ή κυρώσεις για κράτη τα οποία δεν τηρούν τις δεσμεύσεις τους και δεν εκπληρώνουν τι υποχρεώσει του. Και αυτό είναι απαραίτητο αν θέλουμε να σημειώσουμε πρόταση παγκόσμιο για την καταπολέμηση παράνομη αλεία. Ε, πρόταση επίση παγκόσμια πιστοποίηση για τα αλλιεύματα. ή ενισχυμένη παγκόσμια συνεργασία για τη διερεύνηση εγκληματικών δραστηριοτήτων. στο πλαίσιο και της ε, σύμβασης ε, για την καταπολέμηση ε, των ναρκωτικών και του εγκλήματος της διατλαντικής αυτής σύμβασης που δημοσιεύθηκε την Άνοιξη και νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία. Επίσης, ο λεγόμενος συνασπισμός των προθήμων, συμμαχία των προθήμων, που θα μπορούσαν να κάνουν κάτι μαζί. Ξέρουμε ότι στον παγκόσμιο στίβο, στο ΦΑΟ, και στους RFMOs, ε, στους περιφερειακούς οργανισμούς. Ε, γίνονται κάποια πράγματα και καλό θα ήταν να κάνουμε από κοινού ε, πρόοδο. Δεν ξέρω τι πιστεύουν οι εκπρόσωποι της ε, Ιαπωνίας και τον ΗΠΑ, αν θεωρούν ότι πρέπει να προχωρήσουμε με την νομοθεσία περί παρανομισσαλίας και αν πρέπει να υπάρχει κάποιος συντονισμός. Αν μου επιτρέπει, Πρόεδρος, θα ήθελα να προτείνω το εξής. Να ακούσουμε καταρχάς τους ομιλητές από τις αντιπροσωπείες και εν συνεχεία να ξαναπάρω εγώ το λόγο και να σας παρουσιάσω τις ε, τροπολογίες που προτίθεμαι να υποβάλω για την έκθεσή μου. Αλλά αυτό αφού ολοκληρώσουμε τη συζήτηση με τους εμπειρογνώμονες. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ κυρία Λέβιν. Ας μην καθυστερούμε άλλο, θα δώσω αμέσως το λόγο στην πρώτη λύτρια, την κυρία Ρεμπέκα Λέντ. Την ε, σύστησε η κυρία Λέβιν, οπότε δεν χρειάζεται να επαναλάβω την ιδιότητά στο πλαίσιο της Αμερικανικής κυβέρνησης. Έχετε το λόγο κυρία Λέντ για να μας κάνετε την παρουσίασή σας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε και οι Ηνωμένε Πολιτείε πιστεύουν ότι η σωστή ε, εφαρμογή ε, είναι βασική και ε, ε, σε αυτό το σημείο θα ε, σας δείξω τι κάνουμε στις Ηνωμένε για να μπορέσουμε να επιλύσουμε αυτό το θέμα διότι 25% των προϊόντων ε, αλλιεύονται παρανόμως υπάρχουν πάρα πολλά είδη ε, πλοίων που ασχολούνται με την αλληλεία και ουσιαστικά ε, πρέπει να μπορέσουμε αποτελεσματικά να διαχειριστούμε τους πόρους μας και πρέπει να προσπαθήσουμε να τα προχωρήσουμε. Ε, οπότε υπάρχουν πάρα πολλές ε, χώρες, ε, πάρα πολλές περιοχές ή στις Ηνωμένε Πολιτείες και είτε οι Ηνωμένε Πολιτείε είτε σαν κράτος σημαίας είτε σαν κράτος λιμανιού παρακολουθούν τα συστήματα προσπαθώντας να διαχειριστούν σωστά και το οικολογικό σύστημα και ε, υπάρχει μία διαφορά βέβαια μεταξύ της νομιμότητος και της βιωσιμότητος. Μπορεί να έχουμε βιώσιμες μεθόδους που δεν ε, είναι αποδεκτές και βιώσιμες και το αντίστροφο. Υπάρχει όμως συνήθως ε, μία διασύνδεση μεταξύ της παρανομίας και της μη βιωσιμότητος ε, ε, βλέπουμε ότι υπάρχει ε, ένα μια ευρία περιοχή όπου αλλιεύουμε στις Ηνωμένε Πολιτείες και επιπλέον υπάρχουν πάρα πολλοί υπεύθυνοι οι οποίοι παρακολουθούν από ξηράς υπάρχουν δικηγόροι οι οποίοι προβαίνουν στη δίωξη των παραβατών και πλέον αυτού υπεύθυνοι για την εφαρμογή της νομοθεσίας στα κρατικά ύδατα, στα χωρικά ύδατα και επιπλέον δικαστικές αρχές οι οποίες προβαίνουν στη δίωξη. Θα ήθελα να αναφέρω εδώ τον κύριο Στίβενς ο οποίος είναι αυτός ο οποίος παρακολουθεί καταρχήν το σύστημα αυτό ε, οι δυνατότητες ε, εφαρμογής της νομοθεσίας επί του θέματος στις Ηνωμένες Πολιτείες ε, ε, αναλαμβάνονται από την ακτοφυλακή με δύο μικρά πλοία και 57 αξιωματικούς για την, τις παράκτιες δραστηριότητες πλέον αυτών οι οποίες ε, αναλαμβάνονται σε ανοιχτή θάλασσα ε, το βασικό που μας ενδιαφέρει είναι ότι ε, ότι παράνομες δραστηριότητες διεθνώς είναι και στις Ηνωμένε Πολιτείε. Παραδείγματος χάρη η αλληλεία του Αστακού στην Καραϊβική. Ε, μπορέσαμε ε, εφόσον καταλήγουν τα λιεύματα αυτά στις Ηνωμένε Πολιτείε να συνεργαστούμε με γης και ε, να διώξουμε τους υπευθύνους εκ των οποίων μία σειρά κατέληξε στη φυλακή. Επίσης πέραν αυτού σε μία άλλη περίπτωση συνεργαστήκαμε με τους ομολόγους μας στη Νότιο Αφρική και ε, είδαμε ότι ε, ένα μεγάλο μέρος ε, των χρημάτων χρησιμοποιήθηκαν ή στις Ηνωμένε Πολιτείε για να μπορέσουν να να μπορέσει να προχωρήσει το σύστημα είμαστε μεγάλη εισαγωγή και σεβόμαστε το ρόλο μας διότι επηρεάζει και ε, πολλά από τα προϊόντα τα οποία καταλήγουν ε, στις αγορές μας είναι παράνομα αλλιευμένα. Ε, όσον αφορά την αδειοδότηση, προ τεσσάρων ετών είχαμε εστιαστεί στην παράνομη αλληλεία εκτός των χωρικών υδάτων. Παρουσιάσαμε μία έκθεση στο Κογκρέσο. Έχουμε ένα αντίγραφο της εκθέσεως αυτής, εάν σας μας ενδιαφέρει και εντοπίσαμε ε, ποια ε, πλοία ε, διεξάγουν παράνομη αλία και ιδίως τη μη βιώσιμη αλία καρχαρία για να μπορέσουν να αναλυφθούν ενέργειες και να λύσουμε το πρόβλημα υπάρχει μία διοδότηση θετική και πιστοποίηση θετική για αυτούς οι οποίοι έχουν αναλάβει μέτρα και ε, μη θετική πιστοποίηση για αυτούς τους οποίους δεν έλαβαν τα αναγκαία μέτρα. Έξι, είχαν, ε, ε, χώρες είχαν εντοπιστεί, έξι περιπτώσεις στις οποίες αποσύραμε τις άδειες που είχαν χορηγηθεί και ε, σε περιπτώσεις κατασχέσαμε και τα πλοία. Πρόκειται για έξι χώρες όπως είπα και αυτή τη στιγμή ε, διεξάγουμε διαπραγματεύσεις με τις αρχές τους επί του θέματος. Βεβαίως ε, συνεργαζόμαστε και με πολλές περιφερειακές οργανώσεις διαχειρήσεως της αλληλείας και στον κατάλογο λόγω IUU τα, τα ε, εξετάζουμε. Ε, IUU εννοούμε παράνομη λαθρέα άναρχη αλήθεια. Οπότε με τα μέτρα τα οποία έχουμε αναλάβει θα μπορέσουμε ελπίζουμε να διαχειριστούμε την πρόσβαση στα λιμάνια και τον περιορισμό προσβάσεως στα λιμάνια όπου υπάρχουν υπόνοιες Πλέον αυτού οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν ε, διμερή ε, συμφωνία με 46 χρόνια για ε, από κοινού περιπολίες. Έχουμε συνεργασία με τους τους Κινέζους για να παρακολουθούμε την παράνομη αλληλεία στην ανοιχτή θάλασσα και πέραν αυτού τα συστήματα παρακολουθήσεως για, την τελευταία, τα τελευταία 20 χρόνια ενετόπισαν 120 πλοία εκ των οποίων ένα μέρος πλοίων τα οποία παρανόμως εισέρχοντος στα χωρικά μας ύδατα και στα οποία επευλήθησαν κυρώσεις. Οι πολυμερείς συμφωνίες είναι πολύ σημαντικές για να καταπολεμηθεί η παράνομη αλληλεία και θέλουμε ε, να υπάρχουν άδειε εισαγωγής για όλες τις εισαγωγικές εταιρείες. Ε, προσπαθούμε ε, να δούμε ε, εάν υπάρχουν παράνομες εισαγωγές αλλιευμάτων από την ε, Λιβύη ε, υπάρχουν διάφορα επιπλέον προγράμματα για τον ειρηνικό επί των οποίων συνεργαζόμαστε όπως είπαμε τους Κινέζους το, η παρακολούθηση λοιπόν αυξάνεται και προβλέπουμε ότι μέχρι το 2012 θα είμαστε ο πρώτος τομέας στις Ηνωμένε Πολιτείε που θα έχει ολοκληρώσει την οικοδόμηση του συστήματος θα παρακολουθούμε την αδειοδότηση και έχουμε επιπλέον ένα πρόγραμμα παρακολουθήσεως των Τσαλίας του τόνου που παρακολουθούμε ψηφιακά πέραν από ε, ε, την έγγραφη καταγραφή. Ε, συνεργαζόμαστε σε πολλούς τομείς με τις υποανάπτυξη χώρες διότι βλέπουμε όλο και περισσότερες περιπτώσεις εισαγωγών από νότο προς βορρά και αυτή τη στιγμή εντοπιζόμαστε στην Καραϊβική, στη Λατινική Αμερική ε, στο τρίγωνο μεταξύ Νοτιού Αμερικής και Δυτικής Αφρικής και έχουμε προγράμματα παρακολουθήσεως κατά τρόπον ώστε οι χώρες αυτές να έχουν επαρκώς εκπαιδευμένους παρατηρητές πάνω στα πλοία και ε, με αυτά ε, κυρίες και κύριοι σας ευχαριστώ για την ε, ευκαιρία που μου δώσατε να μπορέσουμε να συζητήσουμε μπορέσαμε έτσι να διαπιστώσουμε ότι υπάρχει ανάκληση στο και αδειών από πλοία τα οποία παραβιάζουν την νομοθεσία και ελπίζουμε ότι στη συνέχεια θα υπάρξει μία πιο επίσημη μέθοδος ανταλλαγής πληροφοριών ότι θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τα μέτρα που άπτονται των κρατών λιμένων και να προχωρήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Λέντ. Θα δώσω τώρα τον λόγο στον κύριο Μιαχάρα για να μας κάνει και αυτό τη δική του παρουσίαση και εν συνεχεία θα ξεκινήσει η συζήτηση.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 Καταρχήν επιτρέψτε μου να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς ε, εσάς και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για το ότι μετά το ατύχημα και το παλαιοροϊκό κύμα εξέφρασε τη συμπάθειά της προς τον Ιαπωνικό λαό. Είμαστε πάρα πολύ δύσκολοι και εκτιμούμε ιδιαίτερα την υποστήριξή σας. Θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που μου προσφέρει προσφέρετε ευκαιρία να σας μιλήσω για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία είναι σύμμαχοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια και συνεργαζόμαστε σχεδόν ε, σε όλους τους οργανισμούς ε, διαχείρισης. Έχουμε πάρα πολλά συμφέροντα κοινά που μας ενώνουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ιαπωνία. Ε, έχουμε δεσμευτεί για τη βιωσιμότητα των ελληνικών πόρων. Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία έχουν να επιδείξουν μακρά ιστορία της διαχείρισης των αλληλευτικών πόρων. Μερικές φορές βέβαια έχουμε δύσκολους ε, γείτονες. Εσείς έχετε τις μεσογειακές χώρες, εμείς ε, Έχουμε προβληματικές όμορες χώρες όπως τη Βόρεια Κορέα, την Κορέα, την Κίνα και την Ταϊβάν. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο ε, συνεργαζόμαστε σε πάρα πολλούς ε, τομείς και πιο συγκεκριμένα Υπάρχει φόρουμ συνεργασίας. Γι' αυτό λοιπόν ε, χαίρομαι που μας μου προσφέρει την ευκαιρία ε, να σας απευθύνω το λόγο. Καταρχήν, ε, θα ήθελα να υπογραμμίσω τη σημασία των αγορών. Ε, νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να είναι η πιο σημαντική αγορά για την Αλία. Το 2008 η Ευρωπαϊκή Ένωση εισήγαγε 10 τόνους ψαριών που είναι εντυπωσιακό το, ο αριθμός αυτός. 3 εκατομμύρια η Ιαπωνία, η Κίνα περίπου το, το ίδιο ποσό και στις Ηνωμένες Πολιτείες λιγότερο από 2 εκατομμύρια τόνους. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντική είναι η ευρωπαϊκή αγορά. Το σύνολο της ε, ευρωπαϊκής αγοράς είναι, η ευρωπαϊκή αγορά είναι σημαντικότερος παίκτη ανά τον κόσμο. Αν δούμε λοιπόν το μέγεθος της ευρωπαϊκής αγοράς, πολύ εύκολα κατανοούμε πόσο καινοτόμες είναι οι ρυθμίσεις που εισήγαγε η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της πολιτικής ε, IUU, της παράνομης λατρείας και άναρχης αλίας, IUU όπως θα την αποκαλούμε τώρα στην διάρκεια της ομιλίας. Στην περίπτωση λοιπόν της ε, Ιαπωνίας Έχουμε αυστηρούς νόμους ε, για την διατήρηση του τόνου. Πριν από 15 περίπου χρόνια ε, το κοινοβούλιο μας ε, θέσπισε ένα νόμο για τη διατήρηση του τόνου και με βάση αυτόν τον νόμο ο Υπουργός Αλίας και Γεωργίας μπορεί να επιβάλλει στους αγοραστές και στους εισαγωγείς να καταθέσουν σημαντικές πληροφορίες για τη διατήρηση του τόνου. Εμείς λοιπόν ε, διορθώσαμε πολλά στοιχεία που είχαμε κατά παρελθόν με βάση τη θέσπιση του νέου νόμου. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλές δραστηριότητες που αναπτύσσουμε ως Ιαπωνία, πολλές γειτονικές χώρες και αμφισβητούμενες ζώνες στη θάλασσα που περιβάλλει την Ιαπωνία. Εμείς αντιμετωπίζουμε ε, το πρόβλημα της παράνομης αλίας από τα σκάφη της Κορέας σε ζώνες που ανήκουν στην αλία. Όσον αφορά τον ε, ε, τόνο, τον ερυθρό τόνο, για μας ε, εκεί εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα. Ένα άλλο θέμα είναι ε, ότι η Ταϊβάν αναπτύσσει και δραστηριότητες ε, που αφορούν τους καρχαρίες και παίρνουν μόνο το γόνο από τους καρχαρίες και τα απορρίμματα τα ρίχνουν στη θάλασσα γιατί δεν έχουν την δυνατότητα να διατηρήσουν τα ψάρια, τα μεγάλα ψάρια. Παίρνουν τα πτερίγια των ε, καρχαριών και το υπόλοιπο ε, το ρίχνουν στη θάλασσα. Είναι λοιπόν πάρα πολύ δύσκολο για τους Ιάπωνες ε, να εφαρμόσουν τους νόμους ε, στις εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανοιχτή θάλασσα ε, δεν είναι το σημαντική για μας. Η ανοιχτή θάλασσα χρησιμοποιείται ως ε, βάση για τις αλληλευτικές δραστηριότητες. Βλέπετε ότι κάθε χρόνο προσπαθούμε να ενισχύσουμε τις αλληλευτικές δραστηριότητες γύρω από την Ιαπωνία. Θα ήθελα να μιλήσω για τους ε, πόρους ε, τόνου και θα ήθελα να σας παρουσιάσω δύο ιστορίες που αφορούν ε, το πώς αντιμετωπίζουμε αυτήν την αγορά του τόνου. Βεβαίως και η αγορά της Ιαπωνίας είναι πολύ μεγάλη και βλέπετε ότι καταναλώνουμε μεγάλες ε, ποσότητες ε, ερυθρού τόνου και άλλες άλλα τόνου και μιλάμε για μια πολύ μεγάλη αγορά. Είμαστε ε, πολύ μεγάλη αγορά για σασίμι και κυρίως όσον αφορά τον ερυθρό τόνο καταναλώνουμε το 80% ερυθρού τόνου στον κόσμο. Βλέπετε ότι και πολλές μεσογειακές χώρες εμπλέκονται ε, στο εμπόριο του ερυθρού τόνου. Και έχω λοιπόν δύο ιστορίες, μία επιτυχημένη για την αλία τόνη, μία επιτυχημένη, η άλλη ε, αποτυχημένη. Η πρώτη αφορά τα παραγάδια. εντοπίσαμε πολλά σκάφη πριν από 10 χρόνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και μετά από ε, τρία χρόνια ερευνών που έγιναν στο πλαίσιο του νόμου διατήρησης ε, του τόνου συγκεντρώσαμε πολλές πληροφορίες από τους αγοραστές των προϊόντων ερυθρού τόνου και εντοπίσαμε ε, περίπου 87 αληφτικά σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα αυτά ανήκαν και τα χειριζόντουσαν ε, εταιρείε της ε, Ταϊβάν. Έγινε λοιπόν έρευνες, έγιναν έρευνες για τα σκάφη αυτά Ε, βλέπετε λοιπόν ότι στην περίπτωση του ερθρού τόνου σασίμι η Ιαπωνία έχει τη σημαντικότερη αγορά. Γι' αυτό λοιπόν ε, χρησιμοποίησαμε τα στοιχεία που έχουμε για να περιορίσουμε τις δραστηριότητές τους. Μπορέσαμε λοιπόν να περιορίσουμε σημαντικά τον αριθμό των σκαφών αυτών σε δύο το 2000 και τώρα έχουν εξαφανιστεί σχεδόν όλα τα αλληλευτικά σκάφη τόνου με παραγάδια. Το 2002-2003 τα στατιστικά στοιχεία για την παραγωγή του τόνου επέδειξαν βελτίωση και εμείς βεβαίως ε, ωφεληθήκαμε από αυτή την εξέλιξη. Γι' αυτό λοιπόν επισκεπτόμαστε κάθε μήνα την ε, Ταϊβάν ε, για να μπορέσουμε να εποπτεύσουμε στην διάλυση των σκαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να εποπτεύει κανείς στην παράνομη αλία. Αυτό νομίζω είναι το σημαντικότερο διάβασα την έκθεση της Επιτροπής και νομίζω ότι υπάρχουν όλα τα αποτελεσματικά εργαλεία. Παράλληλα όμως θέλω να σας αναφέρω το ότι είναι εξίσου σημαντικό το πώς χρησιμοποιεί κανείς αυτά τα εργαλεία. Πρέπει να έχει μια καλή στρατηγική που να βασίζεται στα απορίσματα της έρευνας και καλείται κανείς και να εντοπίσει ποιος κάνει ακριβώς τι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ε, κυρίως εσείς ε, ε, μπορείτε να διορθώσετε δεδομένα από τους αγοραστές, νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ε, τώρα θα αναφερθώ στον τόνο του Ατλαντικού. Ε, παρακολουθήσαμε ε, τη διαδρομή από την Αλία μέχρι την αγορά και σας ευχαριστούμε που μας ε, βοηθήσετε να έχουμε αυτό το σύστημα της ιχνηλασιμότητας. Εμείς δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά και τώρα νομίζω ότι έχουμε εντοπίσει κάπως ε, την παράνομη αλία. Η επόμενη περίπτωση είναι η εξής. Εδώ δεν πρόκειται για κλασικές δραστηριότητες παράνομης αλίας με την αυστηρή Πρόκειται για τον έλεγχο της επέκτασης των αλληλευτικών δραστηριοτήτων. Θα ήθελα λοιπόν να υπογραμμίσω ακριβώ αυτό το γεγονός. Αφού λοιπόν εντοπίσαμε τα σκάφη που ε, αλεύουν παράνομα με παραγάδια, ε, βλέπουμε ότι οι μηχανότρατες ε, αλλιεύουν ε, μεγάλες ποσότητες ε, τόνου ανά τον χρόνο, ανά, ανά έτος. Οι επιπτώσεις των μηχανότρατων είναι πολύ σημαντικές. Τα χρήματα από την Κίνα χρησιμοποιούνται για να κατασκευαστούν οι μεγάλες ε, μηχανότρατες. Χρησιμοποιούνται ακόμα και κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατασκευή των μηχανότρατων. Έχει επεκταθεί λοιπόν πρόσφατα η ελευτική δραστηριότητα και η επέκτασή της ε, συνεχίζεται. Ξετάσαμε λοιπόν την κατάσταση όπως το κάναμε ε, και στα ε, ελεκτικά σκάφη με παραγάδια. Το πράσινο κομμάτι δείχνει ε, την Ιαπωνέζικη εταιρεία που εμπλέκεται σε αυτήν την αλληλεία, την FCF. Αυτοί οργα... επένδυσαν και στην Ταϊβάν και στην Κίνα και έχουν κατασκευάσει αυτά τα σκάφη. 38 λοιπόν μεγάλες μηχανότρατες βρίσκονται υπό κατασκευή και οι δραστηριότητε ε, της εταιρεία αυτής συνεχίζονται, εξακολουθούν να κατασκευάζουν μηχανότρατες ε, μεγάλων διαστάσεων. Ε, βεβαίως οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία, ίσως και η Κίνα, αυτές είναι οι μεγάλες αγορές για τα προϊόντα που αλλιεύονται από τις μηχανότρατες. Τώρα όμως πρέπει να συνεργαστούμε γιατί αλλιώς θα καταστραφεί ο τόνος ε, σε ολόκληρο τον κόσμο. Θα ήθελα λοιπόν να σας επισημάνω το εξής. Ε, μιλάμε για μεγάλες εταιρείε ε, στην Ταϊλάνδη, επίσης Ιαπωνέζικων συμφερόντων. Πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε αυτήν την δραστηριότητα γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να ελέγξουμε την άναρχη και παράνομη αλία. Καταλήγω λοιπόν στο εξής συμπέρασμα. θα πρέπει να συνεργαστούμε για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε ε, την παράνομη και αναρχιαλία. Αλλιώς η δική σας συνεισφορά βεβαίως και είναι πάρα πολύ σημαντική ε, στην αντιμετώπιση της ε, παράνομης αλίας. Υπάρχουν όλα τα απαραίτητα μέσα. Τώρα το μόνο που απομένει να ε, συζητήσουμε πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Ελπίζω λοιπόν να μπορέσουμε να συνεργαστούμε και στο εγγύς μέλλον να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά την παράνομη και αναρχιαλία. Ίσως πρέπει να εισαγάγουμε και άλλα μέτρα Τέλος, θα ήθελα να πιστήσω την προσοχή σας στην πολύ κακή αγορά που αντιμετωπίζει η αγορά αλίας. Η εταιρεία η FCF, η μεγάλη αυτή εταιρεία, απέριψε τα ε, προϊόντα της ε, Ιαπωνίας μετά ε, το ε, παλαιολογικό κύμα στην Ιαπωνία. Απέριψαν ε, τα ψάρια μας, ακόμα και αυτά ε, που είχαν αληφθεί την προηγούμενη χρονιά. Προσπάθησαν να μας χτυπήσουν, να κλείσουν την αγορά των κονσερβοποιημένων προϊόντων. Εκμεταλλεύτηκαν δηλαδή την περίπτωση του σεισμού και θέλησαν να μας χτυπήσουν πισόπλατα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ίσως και αυτή να απορρίψει τις δικές μας τις εξαγωγές. Προσέξτε όμως ότι πολλοί ε, χρησιμοποιούν της, ε, την περίπτωση του σεισμού για, ως πρόφαση για να επεκτείνουν την αγορά τους. Ε, σας έχω λοιπόν δώσει ένα βίντεο που αφορά σε αυτά τα στοιχεία που σας ανέφερα και ελπίζω εσείς τα προϊόντα της Ιαπωνίας ε, να τα βρείτε ασφαλή, να μην υπάρξουν προβλήματα. Δεν θα πρέπει να φοβάστε ε, τα ψάρια από την Ιαπωνία, συμπεριλαμβανομένου και του τόνου. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν ε, συμφωνείτε θα δώσω καταρχάς το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο κύριος, για να δω ποιος είναι, κύριος Βερτζίν. Θέλει να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή τις παρεμβάσεις ε, των ΙΠΑ και της Ιαπωνίας. Και πραγματικά ε, πρέπει να πω ότι ηρέμησα κάπως, ανακουφίστηκα, γιατί δεν είμαστε μόνοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αγωνιστούμε κατά της άναρχης παράνομης αλίας. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες ε, και άλλοι εταίροι με διαφορετικά μέσα, ίσως διαφορετικές προσεγγίσεις που έχουν να κάνουν, έχουν να κάνουν με τις ιδιαιτερότητες των χωρών τους, αλλά και αυτοί προσπαθούν να καταπολεμήσουν την παράνομη αλεία. Καλό είναι τρεις ε, ε να καταπολεμούμε την παράνομη αλεία. δεν αρκούν αυτοί σε καμία περίπτωση. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση όπου το μεγάλο μέρος των αλλιευμάτων πολλούνται στις διεθνές αγορές ή φτάνουν προς πώληση στις διεθνείς αγορές χωρίς να γνωρίζουμε κατά πόσον τα προϊόντα αυτά αλλιεύτηκαν νομίμως δηλαδή τα κράτη σημαίας που είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο των αληφτικών σκαφών, δεν ξέρουμε αν έχουν κάνει τους ελέγχους ή τελικά θυσίασαν την νομιμότητα των αλημάτων ή αν τα λιμάνια της ε, μεταποίησης ή της μεταφόρτωσης έχουν και αυτά εφαρμόσει τις διαδικασίες ώστε να φτάσουν νόμετα πρώτα στην αγορά. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε να επιτελέσουμε ένα τεράστιο έργο και θα πρέπει να συσπηρωθούμε και να αφιερώσουμε όλη μας την ενέργεια για να σημειώσουμε πρόοδο. Πιστεύουμε ότι μεγάλες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι καταρχάς να υπάρχει ένα σύστημα πιστοποίησης των αλληλευμάτων. Αυτό είναι το πρώτο εργαλείο που θα μας επιτρέψει να εξασφαλίσουμε ότι κάθε κράτος μέλος αναλαμβάνει τις ευθύνες του και ασκεί τις υποχρεώσεις στο πλαίσιο των ελευτικών δραστηριοτήτων και του ελέγχου. Και βέβαια ο ρόλος του κράτους σημαία είναι πολύ σημαντικός. Και η επικαιρότητα ίδια μας καλεί να επιμείνουμε ξέροντας ότι υπάρχουν ε, διάφορες απόπειρες αποσταθεροποίησης του ρόλου του κράτους σημαίας προς όφελος άλλων κρατών που έχουν απλά εμπορικά συμφέροντα σε όλη αυτή την υπόθεση. Πάντως, επαναλαμβάνω ότι είναι ένα τεράστιο ε, έργο αυτό που μας αναμένει. Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε μια προσπάθεια, προώθησε την ιδέα ενός πιστοποιητικού αλλιευμάτων. Γενικότερα έγινε μια προσπάθεια στην περιφερεια, στις περιφερειακές οργανώσεις ε, διαχείρισης αλλίας, αλλά η επιτυχία ήταν πολύ περιορισμένη. Βέβαια είναι πολύ δύσκολο για μια οργάνωση να διαπραγματευτεί αλληλευτικά δικαιώματα, να εγκρίνει, να ελέγξει, να έχει τα ελεγκτικά μέσα. Ίσως λοιπόν η καλύτερη λύση είναι να έχουμε ένα σύστημα σε πολύ πιο γενικό, σε παγκόσμιο επίπεδο, στο πλαίσιο της ΦΑΟ παραδείγματος χάρη. Δηλαδή η συζήτηση να γίνει πιο, σε πιο υψηλό επίπεδο. Ήδη έχουμε κάποια αποτελέσματα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι τώρα προφανές ότι το σύστημα που έχουμε εφαρμόσει μας επιτρέπει να ανακαλύψουμε μαζικές, απα... μαζικές απάτες κατά των κανόνων που έχουν ε, εγκρίνει η υποδά και οι οργανώσεις αυτές, οι ΠΟΔΑ, οι περιφερειακές δηλαδή οι οργανώσεις διαχείρισης και τα συστήματα που έχουν θετήσει ε, μας δημιουργούν κάποιες απορίες για ποιο πρέπει να είναι αυτό που θα δίνει αυτά τα πιστοποιητικά. Και εμείς νομίζουμε ότι η ΦΑΟ πρέπει να είναι αυτή η οργάνωση. Βέβαια, ένας ε, ε στόχο, ένα σκέλο είναι αυτά τα πιστοποιητικά. Το θέμα είναι, έχουν αλληλευθεί τα αλλιεύματα. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν σύνορα στην αλία. Δεν υπάρχουν όρια σε ό,τι αφορά την πρόσβαση δείξεις ε, από πλευρά των αρχών. Αν θέλουμε να πετύχουμε και αν θέλουμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα και τις δυσκολίες, θα πρέπει να προωθήσουμε τη διεθνή συνεργασία. Ήδη με κάποιους από τους εταίρους μας έχουμε αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες. Πρόκειται για πολύ μεγάλη, ε, μεγάλου χρονικού ορίζοντα έργο. Πρέπει να υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη όμως. Δεν μπορούμε να καταφέρουμε να συμφωνήσουμε εάν δεν είμαστε βέβαιοι ότι οι εταίροι μας τηρούν εντελώς αυτούς τους κανόνες του παιχνιδιού. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε πάρα, πολλούς, ε, πάρα πολλές επιτυχίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, δηλαδή δεν έχουμε πείσει πολλές χώρες να σημειώσουν πρόοδο. Ε, δεν μιλώ για τις χώρες Ένωσης, αλλά για χώρες που όπως μία που προσκαλέσαμε σήμερα εδώ και δεν εμφανίστηκε. Υπάρχουν θετικά στοιχεία, αλλά δεν μπορούμε να βασιστούμε και να περιοριστούμε σε αυτά. Θα πρέπει και άλλοι φορεί στο πλαίσιο τη διεθνού συνεργασία να έχουν ε, το ρόλο του. Ο παραδείγματο χάρη, παράκτια κράτη, κράτη λιμένα, κράτη σημαία. Στον ε, τομέα αυτό δεν νομίζω ότι είναι ε, ανάγκη να Εφεύγουμε κάτι εντελώ καινούριο. Αρκεί πολύ απλά να αντιλήσουμε κάποια έμπνευση εκεί που τέθηκαν τα προβλήματα και να δούμε πώς ρυθμίστηκαν εκεί τα προβλήματα. Και θα δούμε ότι αυτό έγινε με την υιοθέτηση μέσων για την υιοθέτηση και την θέσπιση διεθνών συστημάτων με πολύ σαφείς κανόνες, με πρόσβαση στις αποδείξεις και προστασία των αποδείξεων, κάτι που είναι σημαντικό για τους ε, φορείς που δραστηριοποιούνται. Και θα πρέπει όλοι να προσχωρήσουν σε αυτό το σύστημα ώστε να αποφύγουμε. Αν έχουμε λοιπόν κάποιες συνεργασίες μεταξύ των βασικών εταίρων, οι ελευθερικέ δραστηριότητε, όταν γίνονται σε ένα άλλο, σε άλλο κράτος ή όταν έχουμε ένα άλλο κράτος σημαία, αυτό να καταργεί εντελώς αυτή τη δυνατότητα συνεργασίας. Γι' αυτό θεωρώ ότι η μόνη οργάνωση που θα μπορούσε να προωθήσει τέτοιου είδους μέσα και εργαλεία είναι η ΦΑΟ. Πιστοποίηση λοιπόν των αλλιευμάτων, συνεργασία για την ε, αποκάλυψη κάποιων παράνομων δραστηριοτήτων. Καλά είναι αυτά, αλλά δεν αρκούν. Πρέπει να δούμε τι σημαίνει παράνομη αλληλεία. να μην το δούμε μόνο μέσα από τον παραμορφωτικό φακό ε, του μεγέθους του ματιού του δικτυού. Τι είναι η παράνομη αλληλεία ουσίας. Είναι μια δραστηριότητα που ουσιαστικά έχει ως αποτέλεσμα την οικειοποίηση με παράνομα μέσα κάποιου προϊόντος. Πρέπει λοιπόν να χαρακτηριστεί αυτό ως αδίκημα ε, από ποινικής πλευράς. Αν θέλουμε όμως να είμαστε και ρεαλιστές, γιατί πρέπει να είμαστε, ποινικό χαρακτηρισμός ε, τη παράνομη αλληλεία έχει ως αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται ε, και πιο αποτελεσματικές και διευρυμένες μέθοδοι έρευνας που θα δίνουν πρόσβαση σε μηχανισμούς διεθνούς συνεργασία κάτι που βλέπουμε με επιτυχία να γίνεται σε άλλους τομείς και θα επιτρέψει αυτό επίσης να υπάρχει συνεργασία με την καταπολέμηση άλλων μορφών διακίνησης ή λαθρεμπορίου που σχετίζονται συχνά με την παράνομη αλληλεία ή που γίνονται, διαπράττονται σε σχέση ή πάνω σε σκάφη που αλλιεύουν παράνομα. Παραδείγματο χάρη βλέπουμε σχέση παράνομης αλληλεία σε οργανωμένο εγκλήματος. Μόνο εάν ποινικοποιηθούν οι παράνομες αληφτικές δραστηριότητες θα μπορέσουν να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Τώρα, η θεσμοθέτηση νέων εργαλείων καλό είναι, αλλά δεν αρκεί. Μια δραστηριότητα η οποία διέπεται πάνω απ' όλα από εμπορικά και οικονομικά συμφέροντα ε, έχει ως αποτέλεσμα κάποιοι φορείς να μην θέλουν να παίξουν αυτό το παιχνίδι. Άρα καταφεύγουν, να θέλετε, στο κράτος σημαία ή στην προστασία κάποιου άλλου και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί πιστοποίησης και συνεργασίας, χαρακτηρισμού των περιστατικών και των συμβάντων, που θα στηρίζονται όμως από μηχανισμούς εμπορικών κυρώσεων που θα επιβάλλονται σε αυτούς οι οποίοι ε, με δόλο ή αμέλεια δεν συνεργάζονται στη βιώσιμη διαχείριση των ελευτικών πόρων. Όταν όλες αυτές οι προκλήσεις αντιμετωπιστούν, ληφθούν υπόψη τουλάχιστον, και υπάρξει σχετική λύση, μόνο τότε θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε με βιώσιμο τρόπο τα αλληλευτικά αποθέματα που χρειάζονται οι αλληλείς μας. Το σχέδιο έκθεσης περιλαμβάνει πολλές προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Περιορίζω βέβαια εγώ την δική μου παρέμβαση σε λίγους άξονες γιατί θεωρώ ότι αν πετύχουμε πάνω σε αυτούς τους λίγους άξονες θα μπορέσουμε να δώσουμε νόημα και σε όλες τις άλλες προτάσεις της ε, έκθεσης, παραδείγματος χάρη. Επιδόσεις κρατών σημαία ή κρατών λιμένος, επιδόσεις, ποδά. Αυτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους τους ομιλητές. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα λάβω πρώτη το λόγο για να πω τα εξή. Ανεξαρτήτως της ανάγκης ε, δημιουργίας νέων εργαλείων και μέσων ίσως, εγώ νομίζω ότι πρέπει πρώτα απ' όλα να εφαρμόσουμε σωστά τα ήδη φυστάμενα μέσα και εργαλεία που έχουμε στη θέση μα για την καταπολέμηση τη παράνομη. Αλλιώ, όπω είπε και ο κύριο Μιγιαχάρα, τα κράτη τη αγορά έχουν ειδική ευθύνη για την εφαρμογή όλων αυτών των μέτρων. Ο κύριος Μιαχάρα νομίζω ότι πολύ καλά μας τόνισε τι συμβαίνει σε μια ε, περιφερειακή οργάνωση αλληλείας, παραδείγματος χάρη αυτή του Δυτικού Ειρηνικού μας είπε τι είναι αυτά τα οποία δεν πρέπει να γίνονται. Υπάρχουν ε, συμβαλόμενα μέλη, ε, μέρη και βλέπουμε τι γίνεται με την αύξηση των αλλιευτικών δυνατοτήτων των ε, αλλιευτικών κρατών. Έχουμε τη Νέα Γουινέα που είναι η αρμόδια υπεύθυνη για το 90% της αύξησης αυτής. Η Ιαπωνία μάλιστα πρότεινε πέρυσι το πάγωμα της αύξησης αυτών των αλληλευτικών ε, σκαφών και πήγαν στα νησιά Μάρσαλ και είπαν ότι κατασκευάζουν τέσσερα νέα αλληλευτικά σκάφη 20 εκατομμύρια ευρώ αξία στο καθένα. Ποιος είναι πίσω από όλα αυτά στις νήσους Μάρσαλ. Παπουασία, Νέα Γουινέα, μετά ορίεται και αυτή και τα λοιπά. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι υπάρχουν καταστάσεις ανεξέλεγκτες μεταξύ άλλων γιατί υπάρχουν συμβαλόμενα μέρη, Καναδάς, Ιαπωνία, ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και τελικά εμείς είμαστε η μειοψηφία. Δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά περισσότερα. Υπάρχουν και κάποιες άλλες αντιφάσεις δηλαδή, η Παπασία Νέα Γωνία, παραδείγματος χάρη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει ζητήσει παρέκκληση των κανόνων, έχει κάνει μάλλον παρέκκληση με τους κανόνες προέλευσης. Οπότε ανοίγουμε μία αγορά εκεί όχι στην παράνομη λαθρέα αλία όπως γίνεται στην Ισπανία, αλλά ε, σίγουρα μια αλία που θα έχει και κάποιες παράπλευρες ζημίες για τη δική μας παραγωγή και τις δικές μας αγορές κτλ. κτλ. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες αντιφάσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα πολύ καλό εργαλείο τον κανονισμό για την παράνομη λαθρέα δηλωτή αλία. Εκεί λέγεται ξεκάθαρα ότι όσες χώρες είναι σε περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης αλίας, συμβαλόμενα μέρη δηλαδή, που όμως στην πράξη δεν αποδέχονται δύο βασικά μέσα. Το Catch Documentation Scheme και τα Port State Measures δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να εξάγουν σε αγορές όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε την νομοθεσία που θα εμπόδιζε και θα απέτρεπε όλα αυτά, αλλά αυτή η εφαρμοσία δεν τηρείται. Τα εμπορικά μέτρα σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι είναι εντελώς αδύνατο να τα παρακάμψουμε γιατί είναι το μόνος τρόπος να καταλάβουν οι χώρες ότι εδώ μπαίνει μόνο όσοι, ε, μπαίνουν μόνο όσοι τηρούν τις αρχές. Δεν γίνεται να μιλάβουμε αυτά τα μέτρα. Με τις χώρες της αγοράς νομίζω ότι έχουμε μια κοινή ευθύνη, σοβαρή ευθύνη για όσα γίνονται. Θα πρέπει ο ληφτικός μας τόλος να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις ναι, αλλά όλα αυτά τα ζητήματα πρέπει να τα λύσουμε και η έλλειψη πολιτική βούλησης είναι πάρα πολύ σημαντική. Εγώ μιλάω για την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τη ΣΥΠΑ ή για την Ιαπωνία. Εγώ θέλω πρώτα ε, να πω για τα του οίκου μα. Δεν μπορώ να μιλάω για το τι γίνεται αλλού. Ξέρουμε τι γίνεται και με την Κάνα και με άλλες χώρες. Λοιπόν, έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη ε, δυσκολία. Ε, πρέπει να βρούμε την απαραίτητη πολιτική βούληση. Πρέπει οι υφιστάμενοι κανονισμοί που ισχύουν να εφαρμόζονται και μετά να δούμε για νέα μέσα. Δεν εφαρμόζονται όμως οι υφιστάμενοι ε, κανονισμοί. Γιατί τη Western είπατε εσείς και ο κύριος Μιαχάρα ξέρει πολύ καλά τι συμβαίνει. Λοιπόν, τα είπα και ξαλάφρωσα, πήρα πρώτο λόγο να δώσω τώρα ε, σε συναδέλφου ε, το λόγο. Ναι, πράγματι ήσασταν κατηγιστικοί κυρία Πρόεδρε, όπω πάντα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την ε, παράνομη αλληλεία, πράγματι, όπω είπε και ο πρόσωπο τη Κομισιόν, δεν είμαστε μόνοι μα και είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον της για το μέλλον τη κοινωνίας, να βρούμε τις σωστέ ποινικέ και διοικητικέ διαδικασίε για την καταπολέμηση τη μάστιγα αυτή. Σε ό,τι αφορά την κυρία Λέντα, η οποία είπε ότι υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο, είπε ότι υπάρχουν πολλοί οργανισμοί, θέλω να τη ρωτήσω αν δεν απατώμε, 10 έως 25% της παράνομης αλίας, δεν ξέρω ακριβώς ποιο είναι το ποσοστό των εισαγωγών παράνομων αλιευμάτων που ελέγχουν, θα ήθελα να μας πείτε. Μέσα σε πόσα χρόνια καταφέρατε να μειώσετε και να σημειώσετε την ε, επιτυχία που έχετε και ποιος ήταν ο προϋπολογισμός σας και για τον κύριο Μιά Χάρα. Όπως όλες οι χώρες έχετε και εσείς ε, προβλήματα και η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει προβλήματα με γειτονικέ χώρες. Και η Ευρώπη συγκεκριμένα έχει προβλήματα και πολλά μάλιστα. Μιλήσατε για συντονισμό. Θέλω όμως να μας πείτε και για συγκεκριμένα μέτρα. Επίσης, ό,τι αφορά τον ερυθρό τόνο που είστε μεγάλη αγωγή, ε, ποιες επιτυχίες έχετε σημειώσει. Eh, Ευχαριστώ. Ποιος θέλει το λόγο, κυρία Λέβιν. Ευχαριστώ και τις ε, ευχαριστώ όλους τους ομιλητές διότι όντως εάν δείτε τα ε, τα, ε, τους αριθμούς βλέπετε ότι η Ιαπωνία εισάγει το 70% η Ευρωπαϊκή Ένωση το 60% της αλίας που καταναλώνει όλοι βασιζόμαστε στις εισαγωγές έχουμε τεράστια ευθύνη αλλά και δυνατότητα να κάνουμε κάτι για τις αγορές ε, ήθελα λοιπόν να ε, σας ε, ρωτήσω. Μιλήσατε για ένα σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής και αναγνωρίσεως που οργανώζεται με την Ιαπωνία. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω εάν εσείς μπορείτε να προσυπογράψετε και το σύστημα της ε, παρακολούθησης αλίας. Επίσης πέραν αυτού για το Lacey Act, ε, την νομοθετική διάταξη του Κογκρέσου η οποία λέγει ότι εάν εντοπιστεί παράνομη αλία μπορείτε να φυλακιστείτε. Ε, εάν είναι κάτι το οποίο μπορεί να ε, εμπλέξει την ευθύνη της αγοράς και των λιανοπολιτών. Επίσης, μιλήσατε ε, για τις έρευνες και για τη στρατηγική. Πιστεύω ότι και αυτό είναι κρίσιμο ε, στα πλαίσια αυτά. Και η κυρία Πρόεδρος μίλησε για την πολιτική βούληση και συμφωνώ ότι αν υπάρχει πολιτική βούληση πρέπει να έχουμε εντοπισμένες ε, ενέργειες για να ε, ερευνήσουμε τα, τις ε, περιπτώσεις ε, υπόπτων εγκλημάτων και βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά κράτη με σημαίες ευκαιρίες. Υπάρχουν λοιπόν οι ευθύνες του κράτους της σημαίες αλλά πλέον αυτού υπάρχουν πολλά κράτη τα οποία προσφέρουν σημαίες ευκαιρίες και έτσι δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη. Αυτό είναι κάτι που είναι διεθνώς γνωστό. Η ερώτησή μου είναι τα κράτη της αγοράς ε, τι μπορούν να κάνουν και με ποια συγκεκριμένη στρατηγική μπορούν να αντιμετωπίσουν το συγκεκριμένο πρόβλημα των σημεών ευκαιρίας για τα κράτη σημαίας που δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους πράγμα το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα πολιτικά. Πέραν αυτού, ε, σχετικά με ε, ποιο πιο ανεξάρτητες και τακτικές αξιολογήσεις ε, των επιδόσεων. Η κυρία Ρόμπους έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και εγώ ευχαριστώ τους δύο ε, μυρογνώμονες. θέλω όμως να σας πω ότι λυπούμε πάρα πολύ που δεν υπάρχει κανείς εδώ από την Κίνα διότι θα ήθελα να ακούσω και τις απόψεις που διατυπώνει αυτό το κράτος εσείς πώς πιστεύετε ότι πρέπει να κινηθούμε για να καταπολεμήσουμε την παράνομη αλληλεία. πρέπει να ενισχύσουμε τους τους οργανισμούς μας διεθνώς ή θα πρέπει να αναθέσουμε περισσότερα καθήκαντα στα εθνικά κράτη. Εάν θέλετε ε, να υπάρξει ε, μία πιο ε, μεγάλη ενίσχυση του ποδά, πέστε μου πώς το βλέπετε. Διότι πιστεύω ότι πρέπει να γνωρίζουμε όλα τα στοιχεία και εδώ δεν απευθύνομαι σε εσά προσωπικά, δεν σας προσάπτω κάτι, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει απόκρυψη ορισμένων στοιχείων και ε, λέγει ήδη ότι πρέπει να υπάρξει ποινική δίωξη της παράνομης αλίας. Αναρωτιέμαι λοιπόν πώς θα γίνει αυτό στις ε, διαφορετικές δικονομίες όσον αφορά την ε, αστυνομία, την δικαιοσύνη, τα διάφορα θεσμικά όργανα. Ήδη σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε πολλά προβλήματα. Αναρωτιέμαι λοιπόν πώς αυτό θα οργανωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Είπατε πολύ σωστά ότι τα κράτη ε, που έχουν τις αγορές που διαθέτουν τα προϊόντα θα πρέπει να επέμβουν και αυτό θα πρέπει να παρουσιαστεί. Μπορείτε να μας πείτε συγκεκριμένα πώς πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να γίνει καλύτερα κατά τη γνώμη σας. Δηλαδή, ε, ε, εφόσον είμαστε ένας ισχυρός ομόλογος με 10 εκατομμύρια καταναλωτές, πόσο εσείς διαβλέπετε ότι μπορούμε ε, να προχωρήσουμε προς τους Ιάπωνες συναδέλφους μας. Είπατε ότι υπάρχει κάποια νομοθεσία στη χώρα σας. Πώς οργανώνεστε όμως, πόσους ελεγκτές έχετε, πώς διαχειρίζεστε αυτούς τους ελεγκτές. Εκτός από τον ερυθρό τόνο έχετε και δυνατότητα παρακολουθήσεως άλλων μορφών και επίσης για τον καταναλωτή μας η κατάσταση σχετικά με τη Φοκουσίμα. Πώς έχει εδώ, μιλάμε για παράνομη αλληλεία και πρέπει να προϋποθέσουμε ότι και εκεί θα υπάρχει, σε εκείνη την περιοχή θα υπάρχει παράνομη αλληλεία και ε, την ε, περιοχή μου μόλις είχαμε ένα μεγάλο σκάνδαλο τροφίμων το οποίο δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε ε, είδαμε αν λοιπόν βρούμε ένα ψάρι με υψηλό ποσοστό δηλητηριάσεως πώς θα το παρακολουθήσουμε και πώς αυτό το μολυσμένο προϊόν θα αποφευχθεί να καταλήξει στην αγορά. Και με εδώ μιλάμε για τα ψάρια. Θα ήθελα να κάνω μια επιπλέον ερώτηση στην κυρία Λέντ. Μετά τις ε, τελευταίες πληροφορίες που υπάρχουν για την ετικέτα Dolphin Safe ε, στο πλαίσιο του ΠΟΕ και μετά από όλη τη μάχη που έγινε μεταξύ ημών και του Μεξικό. Τέλο πάντων, το Μεξικό προ εσά. Όποιο ήταν ε, αυτός αυτό που ε, ξεκίνησε την όλη co Eco-labeling, ε, όλα αυτά θα διατηρηθεί αυτό στο μέλλον. Εμένα με ενδιαφέρει γιατί εγώ είμαι ένθερμη υποστηρίκτρια όλων ε, των οικολογικών ε, σημάτων. Τώρα δεν ξέρω ακριβώ με τον Dolphin Safe, αλλά τέλο πάντων, τι έχετε να μα πείτε, μπορούν να διατηρηθούν τέτοιου είδου ετικέτε ε, μετά τα τελευταία, όπω φαίνεται, αποτελέσματα που υπήρξαν στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Κοιτάξτε, Γνωρίζω ότι στις Ηνωμένε Πολιτείε, ε, κατά το παρελθόν υπήρχαν ε, προβλήματα με ΜΚΟ όπως η Earth Island ε, που έχουν τις δικές τους τις ετικέτες φιλικές προς τα αδελφίνια και Παρ' αυτά ε, βλέπουμε ότι εξαφανίζονται ε, ακόμα και καρχαρίες, ε, θαλάσσιες χελώνες. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και η ετικέτα δεν το εξηγεί αυτό στους πολίτες κατά το παρελθόν. Ήταν και απειλητικές αυτές οι ΜΚΟ. Ε, τους είπαν ότι αν δεν χρησιμοποιείτε τα, τη δική μας ετικέτα θα σας βάλουμε σε μαύρη λίστα, σε μαύρο κατάλογο στην ιστοσελίδα μα. Αν λοιπόν ε, κάνει κανείς, ε, λειτουργεί κανείς με αυτόν τον τρόπο, νομίζω ότι δεν είναι αποδεκτό. Λοιπόν, ποιο θέλει το λόγο. Α, όχι, να δώσω κατάρχα το λόγο στην κυρία Λέντ και μετά στον κύριο Μιγιαχάρα. Κυρία Λέντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και όλους σας ε, για τις πολύ ε, ενδιαφέρουσες απαντήσεις που, δώσατε, ε, που θέσατε και ελπίζω να δώσω ικανοποιητικέ απαντήσεις. Καταρχήν όσον αφορά τα αποθέματα, δεν έχω μαζί μου τα στοιχεία. Υπάρχουν πάρα πολλοί φορείς που εμπλέκονται. Μερικές εξ αυτών λειτουργούν ως θαλάσσιοι οργανισμοί. Εν πάση περιπτώσει, εγώ μπορώ να σας δώσω κάποια στατιστικά στοιχεία ως προς τα αποθέματα, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι έχουμε 60.000 προσωπικό, 30.000 βρίσκονται ε, συνεργαζόμενοι κατόπιν τούτου όσον αφορά ε, σε επίπεδο ποσοστών. Είναι πολύ δύσκολο να αναφέρουμε ένα συγκεκριμένο ποσοστό γιατί αν το ξέραμε θα ξέραμε και πού ακριβώ βρίσκεται η παράνομη αλεία. Πάντως στη μασία έχει ότι βλέπουμε να υπάρχει κάποια πρόοδος. Ε, ε, μερικοί βρίσκονται στη φυλακή, επιβάλλονται πρόστιμα. Υπάρχει καλύτερη εφαρμογή τη πολιτική και αυτό είναι πολύ συγκεκριμένο. Κατά τα άλλα είχαμε παράνομα ε, σκάφη της ε, Λιβύης ε, και από τη στιγμή στο ΑΕΚΑΠ μπορούσαμε να επισημάνουμε το γεγονός αυτό, αυτομάτως τους αποσύρθηκε η άδεια. Και στον Παναμά και με εκεί υπήρξαν μέτρα, άρα δηλαδή υπάρχει κάποια πρόοδος. Τώρα, όσον αφορά στην ερώτηση της κυρίας Λουβέν σχετικά με, ένα, με την ύπαρξη ηλεκτρονικού συστήματος. Να πω ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε εργάζονται ε, να υπάρξει ένα ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης για το σύνολο των εισαγών και των εξαγών. Ανεξάρτητα με το ε, πιο ψαριμμένοι, αυτομάτως αναφέρεται στο σύστημα ότι πρέπει να συνοδεύεται από τα εξή παραστατικά και το καθεξής. Αυτό είναι πολύ πιο γρήγορο. Τώρα, όσον αφορά τον ερυθρό τόνο, αυτό πάλι ε, αφορά κυρίως την Ιαπωνία Ίσως ο συνάδελφο από την Ιαπωνία μπορεί να δώσει περισσότερε πληροφορίε. Πάντως η ιδέα είναι ότι αντί να επεκταθεί το γραφειοκρατικό σύστημα, καλύτερα να εστιάσουμε την προσοχή μα στα σημαντικότερα που έχουμε αυτή τη στιγμή, ε, που είναι ε, τα συγκεκριμένα έγγραφα για ε, τον ερυθρό τόνο. Αργότερα, ηλεκτρονικά βέβαια, τα πράγματα θα είναι πολύ πιο εύκολα και γραφειοκρατικά και άλλω πολύ πιο εύκολα να ενταχθούν συγκεκριμένα έγγραφα. Τώρα, όσον αφορά την παράδοση παράνομη αλία εξαρτάται βέβαια από τους πόρου που υπάρχουν και από εκεί εξαρτάται η εφαρμογή συγκεκριμένων προγραμμάτων. Κατά την άποψή μα αυτό που έχει σημασία είναι να έχουμε μια προσέγγιση με βάση τον δεχόμενο κινδύνου. Ε, να ξέρει κανείς ε, τι ε, υπάρχει ε, σε κάποια χώρα που αποτελεί πηγή, αν υπάρχει κίνδυνος, ε, πώς μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά τα περισμένα κονδύλια που έχουμε. Γιατί σε ορισμένε περιπτώσεις δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, πρέπει να έχουμε υπόψη μας το σύνολο του συστήματος και στην εφαρμογή του και να δαπανάμε ανάλογα τα φιντολά κονδύλια. Τώρα, όσον αφορά την νομοθεσία, το θέμα είναι ότι ε, και τα προϊόντα που αγοράζονται πρέπει να ξέρουμε αν είναι όχι και οι παραβάτες να μπουν στη φιλική για κάτι που θα έπρεπε να γνωρίζουν. Ε, προσπαθούμε να ε, πλησιάσουμε τους εισαγωγείς να τους πούμε ότι πρέπει να ξέρετε περισσότερα ας πούμε για τον ερυθρό τόνο από τη Λιβύη τους πήραμε όλους έναν ένα τηλέφωνο που εισήγαγαν ερυθρό τόνο από τη Λιβύη και τους είπαμε προσέξτε γιατί ενδέχεται να βρείτε τον πελά σας που αγοράσατε αυτό το προϊόν νόμος ε, Λέισι ε, είναι πραγματικά αποτελεσματικός και θα πρέπει να εξεταστεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Κίνα δεν ήρθε εδώ, αλλά να πω ότι η Κίνα είναι ένας τεράστιος χώρος εισαγωγών-εξαγωγών και με φθηνό εργατικό κόστος. Ε, τεράστιες εξαγωγές. Ε, εκεί ε, τα προϊόντα μετατρέπονται σε fish sticks και ξαναέρχονται στην Ευρώπη. Πραγματικά λοιπόν λυπάμαι που δεν μπόρεσαν να έρθουν οι συνάδελφοι από την Κίνα. Τώρα όσον αφορά ε, στις πληροφορίες και στα δεδομένα ο κύριος Βερζίν είπε ότι ίσως αυτός πράγματι είναι σωστός δρόμος δηλαδή ανταλλαγή πληροφοριών. Ε, να ξέρουμε τι συμβαίνει με την παράνομη αλία ανά τον κόσμο. Και αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό από το να ξέρουμε μόνο τι συμβαίνει στην αγορά. Όσον αφορά το IDCP, το IDPO, ε, νομίζω εδώ πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν φαντάζομαι ότι θεωρείτε ότι μπορούμε να βρούμε μια λύση. Ο τρόπος με τον οποίο οι ΗΠΑ προσεγγίζουν το θέμα του eco-label, εμείς λέμε αυτό είναι θέμα της αγοράς. Ε, δεν εμπλεκόμεθα, ούτε του καταδικάζουμε αυτές τις ετικέτες, ούτε τις εγκρίνουμε. Απλά προσπαθούμε στους πολίτες μας να δώσουμε όσο δυνατόν περισσότερες πληροφορίες μπορούμε για τα ψάρια και για τη διαχείριση των ψαριών. Στο website μας ε, υπάρχει το Fish Watch. Ε, εκεί μπορεί κανείς να μπει στην ιστοσελίδα και να δει, ας πούμε, παραδείγματος χάνει τάδε ψάρι, ποιος το αλλιεύει, από πού προέρχεται και ούτω καθεξής. Αυτό μπορεί, ας πούμε, να αφορά τον ή οτιδήποτε άλλο. Εμείς δεν καταδικάζουμε ούτε και εγκρίνουμε τις ετικέτες. Το κατά πόσον θα πρέπει να εμπλεκόμεθα σε ε, σκόπιμα παραπλανητικές ε, πληροφορίες, ε, ναι, αν φτάσει κάτι τέτοιο στα αυτά μας, πράγματι εκεί πρέπει να δραστηριοποιηθούμε. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό που πρέπει να κάνουν κυβερνήσεις για το eco-labeling, για τις ετικέτες αυτές, είναι να δίνουν τις απαραίτητες πληροφορίες στους καταναλωτές για να αποφασίζουν μόνοι τους κατά πόσον θα καταναλώσουν το προϊόν ή όχι. Η αλία ε, τα παραλιεύματα, όλα αυτά ε, συνοδεύονται πληροφορίες. Αυτά είχα να σας πω κυρία Πρόεδρε ε, και βεβαίως μετά την συνεδρίασή μας μπορώ και κατηδία να απαντήσω σε ερωτήσεις που ενδεχομένω έχετε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριος Μιαχάρη έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω Καταρχάς να πω ότι κάναμε μια πλήρη έρευνα των δραστηριοτήτων παράνομης ε, αλίας. Χρησιμοποίησαμε όλες τις πληροφορίες που είχαμε από τα τελωνία. Και κάποιες φορές βοήθησε και η αστυνομία. Οι σημαντικότερες πληροφορίες που συγκεντρώσαμε ήταν από τους ομολόγους μας και από εμπορικές εταιρείες. Οι εξαγωγικές χώρες της Ένωσης επίσης μας βοήθησαν και έτσι έχουμε καταφέρει να εκπονήσουμε ένα κατάλογο σε ό,τι αφορά την αλία με παραγάδι. Και μάλιστα δημοσιοποιήσαμε τα αποτελέσματα της έρευνας. Αυτό είναι σημαντικό. Οι μεγάλες λοιπόν εμπορικές εταιρείες, αγοραστές από την ε, Ιαπωνία σταμάτησαν να αγοράζουν προϊόντα από τα σκάφη, από τα πλοία τα οποία είχαν καταγραφεί σε αυτό τον κατάλογο και επίσης δημοσιεύσαμε και ονόματα αγοραστών ε, Ιαπώνων. Οπότε και αυτό ήταν ένα πολύ καλό αποτρεπτικό μέσο. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει διαφάνεια. Αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά τις ε, δραστηριότητες της παράνομης αλίας. Και ενίοτε αντιμετωπίζουμε τη στεναρή αντίσταση Ιαπωνικών εταιριών. Πάντως το κάναμε Και κάποιο είπε ότι χρειάζεται πολιτική βούληση. Ναι, συμφωνώ, χρειάζεται πολιτική βούληση για όλε τι δραστηριότητε. Και για ε, του φορεί τη αλλοδαπή αλλά και τη ημεδαπή. Όλοι θα πρέπει να συμμετάσχουν. Πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση. Θα πρέπει να υπάρχει και ισχυρή πολιτική υποστήριξη. Αλλιώς αναλαμβάνεις μεγάλο ρίσκο. και εμείς το ρίσκο αυτό το ε, αναλάβαμε. Αλλά είχαμε και την ε, στήριξη, την απαιτούμενη. Σε ό,τι αφορά ε, την ε, αναθεώρηση των επιδόσεων πράγματι για όλες τις ποδά χρειάζεται αυτό και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς πρέπει να βοηθήσουν. διάφοροι οργανισμοί όπως η ICAT ε, παράγουν ε, ε, ψηφίσματα, έγγραφα. Η συμμόρφωση όμως δεν είναι πολύ καλή. Πρέπει λοιπόν να ενισχυθεί η συμμόρφωση και να συνοδευτεί βέβαια και από την αξιολόγηση των επιδόσεων. Αυτό είναι το κλειδί για να βελτιώσουμε τις εργασίες μας. Κάποιος ρώτησε ποιος είναι ο ρόλος ε, του RMO. Το ουσιαστικό είναι ότι δίνει κάποιες κατευθύνσεις. Ουσιαστικά οι διμερείς ε, διαπραγματεύσεις είναι αυτές που θα κάνουν τη διαφορά. Αλλιώς οι κανόνες δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Για τις σημαίες ευκαιρίας κάποιος κάτι ε, είπε. Ναι, είναι ένα θέμα αυτό, πραγματικά. πρέπει να δούμε και ποιοι φορείς, ποιοι επιχειρηματικοί φορεί εμπλέκονται. Και πρέπει να δούμε επίσης ε, ποιο κάνει την έρευνα, ε, ποιο ε, αποκομίζει όφελος από διάφορες δραστηριότητες. Πρέπει να υπάρχει συνεργασία, πρέπει να υπάρχει διαφάνεια. Και τότε μπορούμε να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Σε ό,τι αφορά τι γειτονικέ χώρες έχουμε μεγάλο πρόβλημα λαθροθυρία. Και κάποια προϊόντα που έχουν ε, αλλιευθεί λαθρέα επανέρχονται, ε, σε, πηγαίνουν σε κάποιες ε, χώρες που πολύ δύσκολα μπορούμε να ελέγξουμε. Πολύ δύσκολα μπορούμε να ελέγξουμε και να συγκρατήσουμε τις δραστηριότητες αυτές. Η Ρωσία είναι μια εξαίρεση πολλούς, ε, γιατί αλλιεύουν πολλά ε, καβούρια. Υπάρχουν όμως κάποια συστήματα τα οποία έχουν εφαρμόσει και μπορούμε να τα ε, ελέγξουμε αυτά τα παράνομα ρωσικά σκάφη που αλλιεύουν καβούρια. Βέβαια υπάρχουν και άλλες χώρες, Ταϊβάν και άλλοι. Και επίσης υπάρχει πολύ χρήμα που επενδύεται από την Κίνα. Η Κίνα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Υπήρξε πρόβλημα πρόσφατα τουλάχιστον με την Κίνα και πραγματικά πρέπει να έχουμε πολύ σοβαρές ε, συνομιλίες με τις κινέζικες αρχές. Οι επενδύσεις είναι σίγουρα ένας δύσκολος τομέας, αλλά νομίζω ότι πρέπει να δούμε αν γίνονται πουθενά παράνομες επενδύσεις, ε, διότι αλλιώς δεν βλέπω να σημειώνεται πρόοδος αν δεν μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε αυτό το φαινόμενο. Θα ήθελα τώρα να σχολιάσω την ασφάλεια των αλλιευτικών μας ε, προϊόντων σε σχέση δηλαδή με την ραδιενέργεια που μπορεί να έχουν. Πρέπει να σας πω ότι κάνουμε μια ευρύτατη δειγματοληψία κάθε εβδομάδα ε, λαμβάνουμε δείγματα από τα σημαντικότερα ε, αλληλευτικά ε, είδη και άλλα προϊόντα. 100 προϊόντα και παραπάνω ελέγχονται κάθε εβδομάδα. Τα προϊόντα από τη Φουκουσούμα και τις γειτονικές επαρχίες δεν υπάρχει πλέον καμία δραστηριότητα εκεί. Σταμάτησαν μετά τους σεισμούς τα πάντα. Και στη διάρκεια της ελευτικής περίοδου γίνεται δειγματοληψία τουλάχιστον ε, τρεις φορές την εβδομάδα για να μην κυκλοφορήσει στην αγορά κανένα μολυσμένο ψάρι ούτε στην Ιαπωνία ούτε να εξαρθεί προς κάποια άλλη χώρα. Και προσπαθούμε τώρα να εισαγάγουμε μια πλουστευμένη διαδικασία για την αξιολόγηση της ποσότητας ε, της ύπαρξης κάποιας ε, ραδιενεργού ουσίας από το Σεπτέμβριο και μετά θα έχουμε τη δυνατότητα να ελέγχουμε όλα τα αλλιευτικά προϊόντα που ε, φτάνουν ε, στους ε, μεγάλους λιμένες της Ιαπωνίας που είναι και το 95% των συνολικών αλλιευμάτων. Άρα νομίζω ότι θα έχουμε το Σεπτέμβριο και μετά ένα πολύ καλό σύστημα ελέγχου, screening, που γιατί λέω Σεπτέμβριο, γιατί τότε ξεκινάει ουσιαστικά η αλλιευτική περίοδος. Για το Σολομό, Σαρδέλα και όλα τα άλλα αλλιευτικά είδη. Μέρος ε, των αλλιευμάτων εξάγονται και σε άλλες χώρες. Γι' αυτό θέλουμε να φροντίσουμε από τον Σεπτέμβριο και μετά να είναι απόλυτα ασφαλή τα προϊόντα μας. Στο έγγραφο που σας έχω διανύμει θα βρείτε και πάρα πολλές άλλες ε, σχετικές πληροφορίες. Νομίζω ότι αυτά ε, έχω να δώσω σαν απάντηση. Ναι. Ελπίζω να έχω ναι. καλύψει. Κυρία Λέβιν θέλει το λόγο για να κλείσουμε τη συζήτηση. Thank you very much and ε, ευχαριστώ. Ε, όλους τους ομιλητές ήταν πολύ ενδιαφέρον και και θα ήθελα εδώ να συνεχίσω τη συζήτηση για το πόσο μπορεί να προχωρήσουμε και νομίζω ε, είναι πολύ βασικό να έχουμε διμερείς συζητήσεις μεταξύ μας κατά τρόπον ώστε να μπορέσουμε να εντοπίσουμε τις πραγματικές μονάδες, επιχειρηματικές μονάδες οι οποίες εμπλέκονται διότι είναι ε, μια ποινική δραστηριότητα και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε έτσι. Ε, στην ουσία πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε τους βασικούς εμπλεκομένους και να τους αντιμετωπίσουμε. Θα ήθελα εδώ να σας πω τι θα περιλάβω εγώ σαν εισηγήτρια στην έκθεσή μου, σαν βασικά σημεία. Υπάρχει ένα θέμα σχετικά με την ιχνηλασιμότητα. Αυτή η έκθεση μόλις ε, παρουσιάστηκε και πρέπει να ε, αποτελέσει ένα πρώτο βήμα για την ε, βάση δεδομένων σχετικά με το DNA των ε, ψαριών οπότε μπορούμε κατά αυτόν τον τρόπο να γνωρίζουμε τη γεωγραφική περιοχή όπου έχουν αλλιευθεί. Ε, θεωρώ ότι είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε τα διάφορα ψάρια και την παράνομη αλληλεία και θα πρέπει να βρούμε και νέα συστήματα ιχνηλασιμότητος ε, όπως ε, λέχθη και να ερευνήσουμε περαιτέρω το θέμα μία ιδέα ε, ε, που ε, ετέθη σχετικά με το Lacey Act, με την Αμερικανική σχετική νομοθεσία, είναι κάτι που θα πρέπει να εξετάσουμε και στην Ευρώπη, διότι κατά αυτόν τον τρόπο και ο λιανοπολιτής, δηλαδή η άκρη της αλυσίδας της εμπορίας θα μπορεί να φέρει ευθύνη για κατοχή προϊόντων παράνομης είναι κάτι λοιπόν το οποίο θα πρέπει να προχωρήσει και έχω ακόμη να αναφέρω δύο θέματα σχετικά με τις συμφωνίες συνεργασίας των αλλιέων που κάτι που δεν έχουμε επαρκώς αναπτύξει στην έκθεση αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις ε, συμφωνίες συνεργασίας για να ενισχύσουμε την τους περιφερειακούς ελέγχους όπου αναπτύσσονται αυτές τις συμφωνίες. Ήδη έχει εγώ ανέφερα στο δεύτερο σημείο της εκθέσεώς μου το πρόβλημα της ε, ευθύνης αλλά εδώ θέλω να τονίσω την ευθύνη ε, του κράτους της σημαίας και ε, θα πρέπει συγχρόνως να προχωρήσουμε εις τον εντοπισμό των ευθυνών. Εγώ θα τονίσω ότι ευθύνεται το κράτος της σημαίας. Έχω κάνει συζητήσεις με τους χειώδεις εισηγητές και δεν ξέρω αν θα ήθελα να προχωρήσουν και να μας πούν κάτι παραπάνω από αυτού. Διαφορετικά ευχαριστώ την Πρόεδρο. Δεν βλέπω να ζητεί κάποιο το λόγο. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Λέντα και τον κύριο Μιαχάρα που συμμετείχαν στην συζήτηση αυτή. Μία συζήτηση που όπως και κάθε άλλη που έχει να κάνει με την ε, παράνομη λαθρέα και άναρχιαλία είναι ενδιαφέρουσα. Θα τα ξαναπούμε σύντομα στις νέες συνεδριάσεις ε, και της Western και της ε, ICAT και ελπίζουμε να έχουμε τουλάχιστον στο πλαίσιο της Western την απαραίτητη πρόοδο γιατί είναι κάτι πάρα πολύ αναγκαίο. Σας ευχαριστώ. Α, όχι. Πρέπει να αναφέρω και την προθεσμία κατάθεσης ε, τροπολογιών. Α, 20 Ιουνίου το μεσημέρι. Έχει ήδη οριστεί. 20 Ιουνίου λοιπόν. Και έτσι ολοκληρώσαμε με το σημείο 9 της ημερήσιας διάταξης και μπορούμε να περάσουμε τώρα στο σημείο 10. Σύμβαση για τη διατήρηση και διαχείριση των αλλιευτικών πόρων της ανοιχτής θάλασσας στο νότιο ειρηνικό ωκεανό. Η είμαι εγώ. Της προάλλες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μια παρουσίαση της πρότασης. Περί τίνος πρόκειται λοιπόν. οριστικοποίηση λοιπόν ε, για την ε, ζώνη του Νότιου Ειρηνικού που έχει δύο περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης αλίας, την Παναμερικανική Επιτροπή Τροπικού Τόνου και την Western, όπως τη λέμε, την Επιτροπή Αλίας, δηλαδή Δυτικού και Κεντρικού Ειρηνικού, ε, δύο ποδά που έχουν να κάνουν με πάρα πολύ μεταναστευτικά είδη. Ε, θέλουμε να δημιουργηθεί μια νέα ε, πόδα η οποία θα διαχειρίζεται άλλα είδη τα οποία δεν είναι άκρως μεταναστευτικά. Ξεκίνησε η πρωτοβουλία αυτή από τρεις χώρες, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Χιλή, το 2006 με συγκεκριμένα ε, μεταναστευτικά, μάλλον με συγκεκριμένα λευτικά είδη τα οποία θα ρυθμίζονται. τα σαβρίδια και κάποια άλλα βενθικά είδη θα καλύπτονται. Ποιο είναι το κείμενο της ε, σύμβασης. Αυτό το κείμενο εγκρίθηκε το 2009. Εμείς το έχουμε ήδη υπογράψει και τώρα πρέπει πλέον να επικυρωθεί η σύμβαση. Πολύ καλά μας τα είχε πει τις προάλλες ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει να, έχει, να κυρωθεί από 8 τουλάχιστον συμβαλόμενα με τα τρία πρέπει να είναι παράκτια και τα τρία μη παράκτια. Μέχρι στιγμής θα με διορθώσετε αν έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη που δεν γνωρίζω. Το Μπελίζη, Κούβα, η Δανία, ε, της νήσου Κουκ δεν έχουμε κάποιος, νομίζω, ακόμα κάποια εξέλιξη. Οι τρεις χώρες που ξεκίνησαν όλη αυτή την ιστορία, α, με... Λοιπόν, θα έκανα ένα κακόβουλο σχόλιο ότι αυτέ οι τρει χώρε που ξεκίνησαν δύο διαδικασίε δεν έχουν επικυρώσει. Αλλά τελικά από ό,τι βλέπω κάποια ήδη έχει επικυρώσει. Άρα. Άλλο ένα μας λείπει. Ένα τρίτο για να τεθεί σε ισχύ. Θέλω να, και ασκώ κριτική συχνά, αλλά τώρα θέλω να ε, εκφράσω την ικανοποίησή μου. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε μια προσπάθεια ε, σε αυτή την περιφερειακή οργάνωση αλίας να υπάρξει μια διεύρυνση της διαχείρισης των αλλιευμάτων, των αποθεμάτων. Να μην είναι μόνο η ανοιχτή θάλασσα που καλύπτεται. Να καλυφθούν ε, κατά το δυνατόν οι αποκλειστικές οικονομικές ζώνες. Ξέρετε ότι η Σύμβαση της Νέας Υόρκης πολύ ξεκάθαρα ορίζει ότι για τα άκρως μεταναστευτικά είδη οι συστάσεις οι οποίες εγκρίνονται στο πλαίσιο μιας πόδα εφαρμόζονται και στις ε, αποκλειστικές οικονομικές ζώνες αλλά για τα πελαγικά είδη μόνο όταν υπάρχει κάποια συμφωνία για την αλληλεία στην ανοιχτή θάλασσα. Κανονικά πρέπει να εφαρμοστούν όμως παρόμοια μέτρα, παρόμοια μέτρα λέγεται, ε, για τις οικονομικές ζώνες. Προσπάθησε η Κομισιό να δει τι μπορεί να κάνει. Υπήρχαν κάποιες ε, ανησυχίες οι είχαν εκφραστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλαμε να υπάρχει υπεύθυνη οικονομική διαχείριση. Και όταν ήταν δυνατό έγινε αυτή η επέκταση, αυτή η διεύρυνση. Έχουμε τώρα ε, αλλιευτική δραστηριότητα από εννέα ε, κράτη στην περιοχή. Μπελή, Χιλή, Κίνα, Κουκ, Φερόε, Κορέα, Περού, Βανουάτου, Ρωσική Ομοσπονδία. Και βέβαια και Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι την πλήρη έναρξη ισχύω τη σύμβασης Ε, έχει εγκριθεί μια εσωτερική συμφωνία με τον για την αλληλεία πελαγικών ειδών. Έγινε και μια επιστημονική μελέτη την τελευταία ε, χρονιά. Ε, τα σαφρίδια είναι σε πολύ κακή κατάσταση και γι' αυτό πρέπει να υιοθετηθούν κάποια μέτρα. Πρώτα απ' όλα μειώθηκε κατά 40% το ΤΑΚ οι ελευτικές δυνατότητες που χορηγούνται και η ελευτική προσπάθεια επίσης για τα 2007, 2008 και 2009 είδαμε τα σχετικά στοιχεία και είπαμε ότι τα μελλοντικά συμβαλόμενα μέρη θα μπορούν να επιλέξουν ε, ποια είναι η χρονιά που θεωρούν την πιο κατάλληλη για να κάνουν τις ε, προσαρμογές. Πάντως θα ληφθούν ε, μέτρα. Για τα σαφρίδια που είπα είναι το βασικό αντικείμενο αυτής της νέας οργάνωσης διαχείρισης αλίας. Ό,τι αφορά τις αλληλευτικές δυνατότητες είναι 78.600 GT για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Περίπου 10 πλοία ε, αλλιευτικά ε, σκάφη. Μικρή, μικρός είναι μας ε, στόλος κυρίως Ολλανδικά σκάφη αλλιεύουν και είναι και ένα πολωνικό σκάφος. Είχαμε ε, μια συζήτηση, αλλά όταν είχα πάει στην Πολωνία μου είπαν ότι υπάρχει ένα πλοίο πολωνικό που αλλιεύει τώρα. Για, την τον Ευρωπαϊκό Στόλο που είπα είναι κυρίως Ολλανδικός και Πολωνικός, είναι πολύ σημαντική αυτή η αλλιευτική ζώνη για την κατάσταση του σαφριδιού σε άλλους ψαροτόπους ε, που αλλιεύουμε εμείς ε, τα πράγματα δεν είναι πολύ ε, άσχημα. Στο Μαρόκο, παραδείγματο χάρη, στη Μαυριτανία και σε αυτόν τον ψαρότοπο γίνεται η αλλιεύση σαφριδιού κυρίως. Είπα, για να εξασφαλίσουμε το μέλλον του πολωνικού και, και ολλανδικού ελευτικού στόλου που αλλιεύει σαφρίδια σε αυτή την περιοχή, πρέπει να υπάρχει μία να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για να μπορέσουν να συνεχίσουν τι ελευτικέ του δραστηριότητε. Η σύμβαση καταρχήν προβλέπει ότι η Κομισιόν, η Επιτροπή μάλλον, όχι η Κομισιόν, η Επιτροπή εκεί ε, μπορεί να θεσπίσει αλληλευτική προσπάθεια, μέγιστα αλληλευτική προσπάθεια και τάκ για όλη την περιοχή κατανομής του είδους. Υπάρχει κάποιο άνοιγμα. Ε, λέει βέβαια ότι θα μπορεί να καθορίσει. Άρα δεν περιλαμβάνει, δεν ε, περιορίζεται σε αποκλειστικές οικονομικές ζώνες. Το λέει το άρθρο 24. Αν βέβαια με το σύνολο των επιτρεπόμενων αναλυμάτων ή την αλληλευτική προσπάθεια ένα κράτος μέλος δεν συμφωνεί, ένα συμβαλόμενο κράτος, θα μπορούσε να προβάλλει αντιρρήσεις. Επίσης το 25 προβλέπεται ότι μπορεί να ληφθούν επίγοντα μέτρα σε περίπτωση που αναπτύμβαση ε, αλληλευτική δραστηριότητα που ενδέχεται να αποτελεί απειλή για ένα συγκεκριμένο είδο. Η σύμβαση βέβαια τη Νέα Υόρκη για μένα είναι αρκετά παροχημένη, είναι επεπαλωμένη. Δεν έχει να κάνει αυτό τίποτα με, τη, με τα Ηνωμένα Έθνη που δεν νομίζω ότι και ενδιαφέρονται και πολύ για τη δική μου άποψη, αλλά εδώ βλέπω ότι σε σχέση με τη σύμβαση τη, αυτή γίνεται κάποιο άνοιγμα προβλέπεται με αντίρρηση η ένσταση, αλλά μπορεί τα μέτρα αυτά να ε, θεσπίσει η σύμβαση για το σύνολο της ζώνης και όχι μόνο, επαναλαμβάνω, για την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Μια άλλη βελτίωση ακόμα σε σχέση με τις άλλες ε, πόδα είναι η διαχείριση. Ξέρετε ότι η ΝΑΦΟ, η ΆΙΚΑΤ, ε, οποιαδήποτε άλλη η Ισλανδία που δεν είναι κανείς ε, παρούσα εδώ, ε, μπορεί να πει κάποιος ότι ε, βάζω ένσταση για τα τα και τα λοιπά. Και δεν γίνεται τίποτα. Η ΝΑΦΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν κάνει αντίστοιχες αντίστοιχα κατά το παρελθόν. Εδώ όμως υπάρχει κάποιος περιορισμός πλέον. Δηλαδή περιορίζεται η δυνατότητα χρήσης αυτής της διαδικασίας ένστασης ή αντίρρησης. Δεν καταργείται αλλά περιορίζεται. Μπαίνουν κάποιοι περιορισμοί. Και το συμβαλόμενο μέρος που υποβάλλει αυτή την αντίρρηση, αυτή την ένσταση, πρέπει να λάβει εναλλακτικά ισοδύναμα μέτρα. Τουλάχιστον αυτό λέει η σύμβαση. Τώρα θα δούμε πώς θα εφαρμοστούν στην πράξη τα μέτρα αυτά. Αλλά σίγουρα μειώνονται οι λόγια του οποίου μπορεί κανεί να προβάλλει ένσταση και υποχρεώνεται και το συμβαλόμενο μέρο, όπω είπα, να ε, λάβει εναλλακτικά μέτρα αντίστοιχη εμβέλεια. Υπάρχει επίσης ένα για κάποιο σημαντικό ζήτημα που είναι η εγγύηση πρόσβασης ε, στους λιμένες. Με τη χιλή έχουμε ένα θέμα. Υπήρχε απαγόρευση χρήσης των λιμένων της χιλής ε, και για τα πελαγικά ε, σκάφη και για τα θυναλιευτικά. Καταρχήν φαίνεται ότι πλέον εξασφαλίζεται η πρόσβαση στους λιμένες των συμβαλωμένων. Άρα, τα Ολλανδικά για παράδειγμα πλοία θα μπορούν να έχουν πλέον πρόσβαση στη Χιλή. Εγώ ε, θα περιμένω με υπομονησία να δω αν θα το εφαρμόσει αυτό η Χιλή, αλλά έγινε να βήμα προς τα εμπρός. γιατί στο κείμενο, επαναλαμβάνω, εξασφαλίζεται η πρόσβαση των αλληλευτικών πλοίων ενό συμβαλόμενου μέρου στου λιμένε άλλου άλλους συμβαλόμενου κράτου μέλου τη σύμβαση. Καλό θα ήταν ε, να μπορούμε να χρησιμοποιούμε τους λιμένες της Χιλής και όχι του Περού που μιλάμε για 8 ε, μέρες ταξίδι. Λοιπόν, η... ουσιαστικά κάλυψα αυτά τα θέματα. Επαναλαμβάνουμε σας τη διαδικασία λήψεως αποφάσεων και όπως με κάθε ποδά υπάρχει η συνένεση, η διαδικασία της συνένεσης. Αυτός είναι ο γενικός κανόνας. Όταν προβλέπεται ρητά από τη σύμβαση ότι η λήψη αποφάσεων γίνεται με τη συνένεση, υπάρχουν άλλες διαδικασίες που μπορεί αυτό να γίνεται με τα τρία τέταρτα είτε με την πλειοψηφία των μελών. Δηλαδή, για να το πω πιο ξεκάθαρα, ή προβλέπετε ρητά συνένεση ή εκεί που δεν προβλέπετε τρία τέταρτα όταν είναι θέματα ουσίας ή αλλιώς πλειοψηφία. Αυτά είναι τα βασικά θέματα. Δεν ξέρω τώρα αν εκπρόσωποι της Κομισιόν θέλουν να θέσουν κάποιο άλλο θέμα. Εγώ αυτά που θεωρώ σημαντικότερα τα ανέφερα. Και βέβαια πιστεύω ότι πρέπει να στηρίξουμε την πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και νομίζω ότι πρέπει να εγκρίνουμε την δημιουργία αυτής της νέας Οργάνωσης Διαχείρισης Αλίας για τον Νότιο Ειρηνικό. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά, αν κάποιο θέλει το λόγο, μπορώ βεβαίω να τον δώσω. Και Σέσσαρη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ τους πάντες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να σας ευχαριστήσει για το κείμενό σας το οποίο είναι πλήρες και για την εισαγωγή η οποία αναφέρεται στις ε, ε, βασικές ε, γραμμές αυτής της συμφωνίας που περιλαμβάνει τα βασικά σημεία και επειδή θέλω να συμπληρώσω αυτά που είπα στην προηγούμενη μου ανακοίνωση σε αυτή την αίθουσα θα ήθελα να σας πω ότι και οι ευθύνε των κρατών της σημαίας και των κρατών λιμένος τώρα έχουν περιληφθεί στο κείμενο της συμβάσεως δεν είναι δευτερογενής νομοθεσία αλλά βασική νομοθεσία πράγμα το οποίο αναβαθμίζει την όλη διαδικασία. Θέλω να σας πω ότι επιπλέον η Νέα Ζηλανδία κύρωσε την 1η Ιουνίου πέρυσι οπότε μία από τις ε, τρεις χώρες που ξεκίνησαν αυτή τη διαδικασία έχει ξεκινήσει να λειτουργεί συγκεκριμένα Υπάρχει, υπάρχουν μερικά παράκτια κράτη, τουλάχιστον ένα κράτη, παράκτιο κράτος. Έχουμε την Ίσου αλλά χρειαζόμαστε ακόμη ένα και ε, για να προχωρήσουμε και γι' αυτό θέλουμε να ολοκληρώσουμε την ε, κύρωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και για τη την εικόνα που δίνομαι και, για τον ρόλο κατά τις διαπραγματεύσεις. Είναι μια διαδικασία τέτραετής η οποία αντικατοπτρίζει τις βασικές πρόοδους στην νομοθεσία που άπτεται της αλληλείας. Ευχαριστώ. Εάν κανείς άλλος δεν ζητά το λόγο... Έχω ήδη στείλει προς μετάφραση το κείμενο που φαντάζομαι ότι το έχετε και για να δούμε πρέπει να ορίσω προθεσμία κατάσταση τροπολογιών. Ναι, 20 Ιουνίου το μεσημέρι και για αυτήν την έκθεση. Θα ψηφίσουμε τον Ιούλιο στην Επιτροπή μας και θα πάει στην Ολομέλεια την 1η του Σεπτεμβρίου. Καλό είναι λοιπόν να δώσουμε το πράσινο φως ώστε να εγκυρωθεί η σύμβαση το πρασινο φως ωστε να κυρωθει δυνατόν. Κύριε Τσέσσαρ, σας ευχαριστούμε πολύ και δεν νομίζω να υπάρξει κανένα πρόβλημα με αυτό το θέμα. Και μπορούμε τώρα να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, ε, που είναι το σημείο 11. Ο κύριος που έπρεπε να είναι εδώ δεν είναι από ό,τι φαίνεται. Άρα θα περάσουμε στο επόμενο σημείο. Έκθεση του κύριου Βαλίση για την Πολωνία. Λοιπόν, Αφήνουμε το 11 για λίγο αργότερα και περνάμε στο σημείο 12 που είναι η έκθεση για την αποστολή της Αντιπροσωπείας Επιτροπής Αλίας από 18 έως 20 Μαΐου στο Γκτάνσκ της Πολωνίας. Έτσι δεν είναι. Α, κύριε Φερέιρα, θέλατε το λόγο. Το θέμα αυτό θα το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Ε, όχι, αλλά δεν είναι εδώ ο υπεύθυνο της Επιτροπής ο οποίος ε, θα το παρουσίασε, οπότε θα το συζητήσουμε αργότερα. Αν δεν ε, έρθει μόνο τότε θα αναβληθεί. Απλά το αναβάλουμε ενώ το αφήνουμε για μετά, όχι ότι το, το καθυστερήσαμε. Προηγείται το 12 και θα συντομεύσουμε έτσι. Ο κύριος Βαλέσα λοιπόν. Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την επίσκεψη. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, κατά την άποψή μου. Και θα σας δώσω το λόγο. Α, βλέπω ότι ήρθε και ο κύριος Ράμπο, που θα μας ε, ε, αναφέρει τα περί του 11. Λοιπόν, πείτε μας σύντομα, σύντομα την, ε, τι έγινε στην Πολωνία. Ευχαριστώ. E, θέλω να συζητήσω, δεν θέλω να συζητήσω την έκθεση, την έχετε στο φάκελό σας αλλά θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εκπροσώπους της γραμματείας μας οι οποίοι με βοήθησαν να οργανώσουμε αυτή την επίσκεψη. Ελπίζω ότι θα μπορέσω να σας δείξω ποια, ε, ότι μπόρεσα να σας δείξω ποια είναι τα προβλήματα της πολωνικής αλληλείας και ελπίζω ότι σας άρεσε και η χώρα μου και θα θελήσετε να ξαναεπισκεφθείτε την ωραία χώρα μας και ιδίως την στην πόλη μου το Γκτάνσκ που προσπαθεί να γίνει Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα το 2016 και ότι θα μπορέσουμε να ξανασυζητήσουμε τα θέματα της Αλίας. Ευχαριστώ. Έχουμε στείλει και στην, ε, σύμβαση το, στην ε, διάσκεψη των πρώτων επιτροπών ε, την αναφορά μας για να γνωρίζουν τι κάνει η αντιπροσωπεία μας όταν ταξιδεύει στο εξωτερικό. Και τώρα περνάμε στο σημείο 11. Παρουσίασε από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Αγορών Προϊόντων Αλίας και Ιδατοκαλλιέργεια, ΕΜΟΦΑΠ. Μα ήρθε ο κύριο Ρούμπο εδώ πέρα να μας κάνει την παρουσίαση. Καλώ ήρθατε και όταν καθίσετε και βολευτείτε θα σας δώσω το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ που μας δίνετε αυτή τη δυνατότητα σε λίγα λεπτά να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε μία έκθεση σχετικά με την εξέλιξη αυτής της προκαταρκτικής δράσης που ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επέτρεψε να δεσμεύσουμε ε, πόρους για να μπορέσει να ξεκινήσει το πρόγραμμα αυτό. Το πλαίσιο, το πλαίσιο μόλις σας το περιέγραψα ε, προς υπενθύμηση και αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι αυτή η σύμβαση η οποία ξεκίνησε γέρος θα επεκταθεί επί σειρά ετών και θα κατανεμηθεί σε τρεις φάσεις. Καταρχήν θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης και να σας περιγράψω τι θα γίνει στην επόμενη διετία. Ε, σας υπενθυμίζω ότι ο στόχος αυτού του προγράμματος ε, απέβλεπε στον επιτραπή επιτραπεί στους ενδιαφερομένους από την ε, αλία και την υδατοκαλλιέργεια να παρακολουθούν όλη την αλυσίδα κατά τρόπον ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι από πλευράς βιομηχανικής αλλά ε, και πολιτικοί που λαμβάνουν αποφάσεις να μπορέσουν να καταλήξουν ε, σε επικοδομητικές αποφάσεις. Έχουμε δηλαδή μία γενική εικόνα της αγοράς αλίας και υδατοκαλλιέργειας ε, στην Ευρώπη η οποία είναι η πρώτη αγορά ανά τον κόσμο να συγκρίνουμε τις εθνικές ε, αγορές ε, μεταξύ τους, μεταξύ των κρατών μελών και να διαπιστώσουμε την οικονομική κατάσταση της αγοράς αυτής σε σχέση με τη διεθνή αγορά υπενθυμίζοντας ότι πέραν του 65% των προμηθειών μας εξαρτάται από τις εισαγωγές. Ένα άλλο βασικό στοιχείο για να κατανοήσουμε αυτό το πρόγραμμα, τουλάχιστον όπως απορρέει από τις εργασίες οι οποίες αναπτύχθηκαν πέρυσι στην πρώτη φάση, είναι ότι αν θέλουμε ένα παρατηρητήριο έτσι όπως έχει διατυπωθεί στις επιθυμίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δηλαδή για να έχουμε οικονομικές πληροφορίες, για να αντιληφθούμε καλύτερα πώς διαμορφώνονται οι τιμές και τα περιθώρια κέρδους, θα πρέπει το περιθώριο αυτό όχι μόνο να κατανοήσει ε, και να συγκεντρώσει αλλά να αναλύσει όλες τις πληροφορίες σε όλο το μήκος της αλυσίδας και στο πνεύμα αυτό διεξήχθησαν και οι εργασίες μας επίσης πρέπει να υπενθυμίσουμε την κάλυψη αυτού του παρατηρητηρίου το οποίο λαμβάνει υπόψη τρία επίπεδα καταρχήν για να απαντήσω εις ε, την ερώτηση η οποία είχε προκύψει όταν μιλήσαμε για την ανακύωση και την κρίση των καυσίμων είναι να γνωρίσουμε όλες τις πληροφορίες της εσωτερικής αγοράς σχετικά με την αλία και την υδατοκαλλιέργεια και αυτό με τις διακοιμάνσεις οι οποίες έχουν διαπιστωθεί μεταξύ κρατών μελών και θα δείτε αργότερα τα αποτελέσματα. Το δεύτερο ήταν να έχουμε διεθνείς πληροφορίες λόγω της μεγάλης εξάρτησης της ε, αγοράς μας από την διεθνή αγορά. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε συγκεκριμένα ε, ε, τα προϊόντα αυτά. Και τρίτον, Μία βασική πηγή ε, προμηθειών είναι η Ισλανδία και η Νορβηγία οι οποίες είναι ε, μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και ε, επιπλέον με τις χώρες αυτές συμμεριζόμαστε διάφορους φακέλους στα θέματα της αλίας και της υδατοκαλλιέργειας και γι' αυτό ήταν βασικό να γνωρίζουμε αυτή την αγορά. Επιπλέον κατά αυτήν την πρώτη φάση ε, καθορίσαμε τις ε, ε, συχνότητες και το είδος των πληροφοριών που θέλαμε να επεξεργαστούμε. Για να έχουμε την καλύτερη οικονομική απόδοση έπρεπε να καθορίσουμε τη συχνότητα των δεδομένων και τη φύση των δεδομένων ε, ε, στο πρώτο τετράγωνο λοιπόν βλέπουμε τους δικτές ε, τους οποίους λαμβάνουμε υπόψη και οι οποίοι, θα εξετάζονται εβδομαδιαία. Το ενδιαφέρον αυτής της παρουσίασης ή αυτής της εβδομαδιαίας παρακολούθησης είναι να δίνει επαρκείς ε, πληροφορίες στους οικονομικούς παράγοντες όσον αφορά τις εξελίξεις. Το δεύτερο επίπεδο είναι να παρακολουθούμε τις τάσεις της αγοράς και εκεί δεν μιλάμε πλέον για εβδομαδιαία παρακολούθηση αλλά μηνιαία για να χρησιμοποιούμε τις εβδομαδιαίες πληροφορίες και για να μην εστιαζόμαστε σε ορισμένα είδη τα οποία μπορεί κάποια στιγμή του χρόνου να ε, υπάρξουν θύματα μιας κρίσης και να έχουμε μια πιο διαρθρωμένη, καλύτερα διαρθρωμένη ε, δομή και τέλος ε, να υπάρχει ένα τρίτο επίπεδο που θα βασίζεται σε ετήσιες πληροφορίες και θα μας δίνει ε, μία καλύτερη ενημέρωση, ένα καλύτερο πλαίσιο το οποίο θα επιτρέψει εις του, αυτούς που λαμβάνουν τις πολιτικές αποφάσεις να είναι συγκεκριμένοι και να μπορούν να επιλύουν κατά περίπτωση τα προβλήματα της αγοράς αλληλείας και υδατοκαλλιέργειας. Και τέλος όλες οι πληροφορίες οι οποίες ε, μπορούν να αποκομιθούν δηλαδή χωρίς μια συγκεκριμένη σειρά διότι οι σειρές ε, θα εξαρτώνται από το τι ζητούμε αν θέλουμε προσωμιώσεις αν θέλουμε ε, τρόπους αναλύσεως του κόστους και των περιθωρίων κέρδους και θα βασίζονται στις πληροφορίες τις οποίες έχουμε σε όλα τα επίπεδα και βάσει των δεδομένων τα οποία έχουν επικυρωθεί. Αυτά όσον αφορά την ε, ε, ε, σκέψη μας σχετικά με τις συνέχειες και τον τρόπο λειτουργίας αυτού του παρατηρητηρίου και επιπλέον επειδή αναφέρθηκα στο το θέμα αυτό θα πρέπει να δούμε πώς θα παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα και έχετε εδώ μία σειρά προϊόντων που μπορούν να προσφέρονται Παραδείγματο χάρη αναφέρομαι σε μία τάση των τιμών που μπορεί να βασιστεί σε εβδομαδιαίες πληροφορίες ή να υπάρχει μία παρακολούθηση ε, εξελίξεων της πρώτης πωλήσεως κάποιου είδους ε, της τιμής ε, πωλήσεως, της πρώτης πωλήσεως ή της εξαγωγής κάποιου είδους και όλα αυτά σε συνδυασμό με χρήσιμα σχόλια για να κατανοήσουμε τις, δυναμικές, τις οικονομικές δυναμικές. Είναι απλώς δηλαδή μία σειρά από παραδείγματα που αναφέρω σχετικά με το τι μπορεί να προσφερθεί. Δεν είναι εξαντλητικός ο κανόνα, ο, κατάλογος και δεν είναι μόνο αυτά τα θέματα τα οποία μπορεί να πραγματευτεί αυτό το παρατηρητήριο. Ένα άλλο βασικό στοιχείο και βλέπω εδώ ότι ε, παρέκαμψα ε, μία διαφάνεια είναι ότι στο τέλος αυτών των 18 πρώτων μηνών αναλύσεως καταλήξαμε σε μία διαπίστωση, ε, κατέληξε μία διαπίστωση ο σύμβουλος η ΚΟΖΕΑ ε, και μετά από συναντήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατύπωσε την κατάσταση για τις οικονομικές, τα οικονομικά στοιχεία της υδατοκαλλιέργειας και της ε, ε, αλληλείας και θεωρούμε ότι τα στοιχεία αυτά είναι ικανοποιητικά και ότι υπάρχει μία σωστή ε, χρήση. Η δεύτερη κατηγορία είναι οι πληροφορίες ε, όπου υπάρχουν ε, ε, υπάρχουν δεδομένα σχετικά με την φύση των σειρών που θέλουμε να ακολουθήσουμε για τα στοιχεία που θέλουμε να συλλέξουμε και στα γκρίζα μιλάμε για, σήμερα για ισχύουσες και υπάρχουσες πληροφορίες αλλά όχι με ομοιογενή χαρακτήρα. Θέλουμε λοιπόν να υπάρξει μία ομοιογένεια αλλά πρόκειται συγχρόνως για πληροφορίες οι οποίες είναι διαθέσιμες ε, ε, σε, σε συγκεκριμένο τομέα δηλαδή ε, βλέπουμε τι γίνεται στις πωλήσει στο ε, πληστηριασμό στους διάφορους οργανισμούς δηλαδή να επεξεργαστούμε τα στοιχεία που διατίθενται για να μπορέσουμε να γνωρίσουμε πώς αναπτύσσεται οικονομικά η αλυσίδα και όσον αφορά τώρα τα άσπρα τετράγωνα θεωρούμε ότι τα στοιχεία αυτά ελείπουν αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν Οπότε στο στην, ε, ε, στην ολοκλήρωση αυτής της αξιολογήσεως θέλουμε να λάβουμε υπόψη μας τα εξής ε, κυρία Πρόεδρε να μην δημιουργήσουμε καμία νέα υποχρέωση ε, μέσω της ε, κοινωτικής νομοθεσίας διότι αυτή τη στιγμή η κοινωτική νομοθεσία μας δεσμεύει επαρκώς για να μπορούμε να τροφοδοτήσουμε την οικονομική πληροφόρηση και να κατανοήσουμε αυτόν τον τομέα. Άρα πρέπει να επεξεργαστούμε τις ισχύουσες διατάξεις. Επιπλέον μπορούμε να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες οι οποίες υπάρχουν στις εθνικές διοικήσεις <clears throat> δηλαδή στα ισχύοντα ε, δεδομένα τα οποία ήδη υπάρχουν και εδώ παραδείγματο χάρη να αναφέρουμε στις πληροφορίες σχετικά τις ε, αγορές χονδρικής πωλήσεως αλλά ε, ε, πρέπει να σας πω ότι τέτοιες αγορές υπάρχουν μόνο σε τρεις χώρες την Ισπανία, την Ιταλία και τη Γαλλία και δεν μπορούμε να έχουμε τέτοιες πληροφορίες σε άλλες χώρες όπου δεν υπάρχουν αλλά εκεί μπορούμε, όπου υπάρχουν μπορούμε να τα επεξεργαστούμε πλέον αυτού η τα κράτη-μέλη έχουν πληροφορίες σχετικά με την, ε, τις σημειώσεις ε, των πολίσεων που είναι μια κοινοτική υποχρέωση. Άλλες πηγές είναι οι διεθνείς οργανώσεις για την ε, πληροφόρηση, η ΦΑΟ που δεν είναι τόσο δεσμευμένο για την αλία όσο είναι ας πούμε που επίσης χρησιμοποιείται το Globe Fish και υπάρχουν ιστοσελίδες οι οποίες δεν χαρακτηρίζουν μόνο την ε, κοινότητα αλλά την Νορβηγία και την Ισλανδία που έχουν επίσης ιστοσελίδες με οικονομικές πληροφορίες στον τομέα αυτό. Και τέλος για τις ε, λεπτομερείς αναλύσεις που θέλουμε να κάνουμε θα πρέπει να ανατρέξουμε στα στοιχεία τα οποία συνήθως διατίθενται από ιδιώτες και εδώ δεν θέλω να ε, κάνω διαφήμιση αλλά υπάρχουν διάφοροι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή στα κράτη-μέλη ορισμένες ε, εταιρείες οι οποίες προσφέρουν οικονομικές πληροφορίες είτε μόνο για την αλληλεία είτε και πιο γενικές πληροφορίες που καλύπτουν επίσης την αλληλεία. Αγοράζουμε λοιπόν τα στοιχεία αυτά από αυτούς τους παρόχους πληροφορίες χωριών σας, έκανα μία, σας παρουσίασα μία γενική εικόνα της αξιολογήσεώς μας, της διαθέσεως, ε, της υπάρξεως και της ποιότητος των πληροφοριών που πρέπει να αξιολογηθούν ε, από αυτό το παρατηρητήριο και πέραν των πρασίνων πλευρών που θεωρούνται ε, σαν ικανοποιητικές και ποιοτικές πληροφορίες θα πρέπει στους επόμενους μήνες να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τα τμήματα τα οποία είναι μπλε πάνω στη διαφάνεια είναι δηλαδή μία μακροπρόθεσμη εργασία που θα αναλάβουμε με τα κράτη-μέλη και με όλους τους εμπλεκομένους που μπορούν να μας δώσουν τέτοιες πληροφορίες διότι η ιδέα είναι όλοι να συμμετέχουν ή και ο θελός. Ε, πρέπει λοιπόν ότι, ε, να πούμε ότι η ε, επιτυχία της προσπαθίας θα εξαρτηθεί από το εάν θα μπορούμε όντως να εξαρτηθούμε εξυπηρετήσουμε όλους τους ενδιαφερομένους. Και στο ΛΕ τμήμα θέλω να κάνω ένα-δυο σχόλια. Είναι κάτι εφικτό. Αλλά αυτό το οποίο μας προβληματίζει είναι τα άσπρα τμήματα, δηλαδή όπου θεωρούμε ότι ίσως δεν χρειάζονται πληροφορίες σχετικά με την πρώτη ε, πώληση των προϊόντων αλίας. Θεωρούμε ότι η πληροφόρηση αυτή δεν είναι αναγκαία και αν είναι αναγκαία θα επέβαλε μία νέα κοινοτική νομοθεσία που υποχρεώνει τους παραγωγούς να μας, της υδατοκαλλιέργειας να μας δίδουν τα σημειώματα απολύσεων που δεν περιλαμβάνεται στην νομοθεσία σήμερα στην κοινότητα. Θέλουμε συγκεκριμένες λοιπόν πληροφορίες όχι μόνο για την πρώτη πώληση αλλά βάσει των πληροφοριών που θα μπορούσαν να μας δώσουν οι υδατοκαλλιεργητές σε σχετικά με τις μηνιαίες τάσεις της αγοράς τους και τις οποίες ενδέχεται να χρειαστούμε για τη χονδρική πώληση όπως σας είπα είναι ένα σύστημα που δεν είναι γενικευμένο και αυτό είναι ο πρώτος λόγος και επιπλέον στα κράτη-μέλη όπου υφίσταται ε, θα είχαν πρόβλημα να αγοράσουμε τα δεδομένα διότι ε, θα έπρεπε να αντιμετωπίσουμε πολύ λεπτές καταστάσεις ε, και οι εβδομαδιαίοι δείκτες επαρκούν για να καταλάβουμε την δυναμική σε αυτό το επίπεδο της αλυσίδας για τις εξαγωγές δεν έχουμε πρόβλημα. Όσον αφορά τώρα την ε, μεταποίηση, δύο είδη πληροφοριών δεν διατίθενται για απλό λόγο και θα πρέπει να τον σεβαστούμε, διότι ε, στις διαβουλεύσεις μας με τον μεταποιητικό τομέα διαπιστώσαμε ότι τα στοιχεία αυτά μπορεί να μην είναι ακριβώς επαγγελματικό μυστικό αλλά πρόκειται για εμπιστευτικά στοιχεία διότι επηρεάζουν την εμπορική στρατηγική του τομέα και πιστεύουμε ότι ε, αυτό ε, το τετραγωνάκι δεν θα το καλύψουμε και ε, θα καλύψουμε στη μεταποίηση τρία επίπεδα που δεν μας προβληματίζουν ε, ε, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα γιατί μπορεί να έχουμε δυσκολία για να συλλέξουμε τα στοιχεία και θα εξαρτηθούμε πάρα πολύ από τη δυνατότητα αγοράς των πληροφοριών από τους κατέχοντες. Πρέπει όμως εδώ να αναφερθώ και στην άποψη των διαφόρων εμπλεκομένων στην όλη διαδικασία. Ερευνήσαμε και διαπιστώσαμε ότι πρέπει να τους βολιδοσκοπήσουμε για να δούμε πώς αυτοί αντιλαμβάνονται αυτή τη διεργασία. Σιγά σιγά λοιπόν τα κράτη-μέλη εκ των οποίων αρκετά ήταν ε, πολύ αρνητικά στο να μας δώσουν πληροφορίες που θα χρησιμοποιόντουσαν σε κοινοτικό επίπεδο σιγά σιγά ακολουθούν την δικιά μας σκέψη και τονίζω αυτή την ε, πληροφορία διότι στην αρχή ήμασταν αρκετά απεσιόδοξοι σχετικά με την υποδοχή που θα είχαμε από τα κράτη-μέλη σχετικά με το παρατηρητήριο αυτό. Τώρα η βιομηχανία ο τομέας της παραγωγής είτε πρόκειται για την βιομηχανία είτε για την υδατοκαλλιέργεια με διαφορετικές τοποθετήσεις μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι προσιλωμένη επιπλέον ή τουλάχιστον έχουν αντιληφθεί την έννοια αυτού του εργαλείου που είναι βασικό και αντελήφθησαν ότι η πληροφόρηση αυτή μπορεί να τους είναι χρήσιμη στην καθημερινή τους εργασία και από τους παραγωγούς δεν αντιμετωπίσαμε προβλήματα από τους μεταποιητές και τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για να λάβουν αυτές τις πληροφορίες ίσως λιγότερο σαφώς από ό,τι στον τομέα της παραγωγής αλλά θα έλεγα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Αντιθέτως, για τη μεταποίηση, για τους λόγους που προανέφερα, είναι μία, υπάρχει μία στάση αναμονής, wait and see και δεν περιμένω να υπάρξει μεγάλη ενθουσιασμός να μας δώσουν πληροφορίες διότι ε, τις πληροφορίες που έχουν προσπαθούν να τις κρατήσουν για τον εαυτό τους. Τι θα γίνει τώρα στο μέλλον. Είμαστε στη φάση 1. Έχουμε ακόμη να καλύψουμε δύο φάσεις. Τη δεύτερη φάση η οποία προβλέπεται για εφέτος και τις αρχές του 2012 και θα μας επιτρέψει μαζί με τον σύμβουλο την Κοζιά να αναπτύξουμε αυτό το εργαλείο όσον αφορά την πληροφορική του διάσταση διότι θα μπορέσουμε να τα αναλύσουμε ε, και στη συνέχεια τα στοιχεία αυτά να διατεθούν και σε σχέση ε, με το την πρώτη διαφάνεια που έδειξα στη φάση αυτή θα γνωρίσουμε καλύτερα τι πληροφορίες μπορεί να δώσει το παρατηρητήριο σε ενδιαφερομένους και τρίτον η τρίτη φάση δεν είναι όπως είπα είναι ε, τα τεστ αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θέλουμε το οργανισμός που λειτουργεί το παρατηρητήριο να μπορέσει να το λειτουργήσει αλλά θέλαμε να τους διαθέσουμε ένα εργοστάσιο με το κλειδί στο χέρι δηλαδή έτοιμο για χρήση Θέλω να σας ευχαριστήσω και πριν κλείσω μια τελευταία παρατήρηση. Η περίληψη της πρώτης φάσεως του προγράμματος θα διατεθεί στο διαδίκτυο και θα ανακοινωθεί σε αυτή την Επιτροπή ε, την επόμενη εβδομάδα. Είναι ένα ογκώδες έγγραφο το οποίο είναι πολύ λεπτομερές και πιστεύω ότι θα απαντήσει σε οποιοδήποτε ερωτήσεις θα έχουν μείνει μέχρι τότε αναπάντητες. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπό. Κύριος Φεραίρα έχει το λόγο. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον, ε, για αυτή την ομιλία. Θα ήθελα και εγώ να κάνω κάποιες ερωτήσεις, αλλά να κάνω και ένα σύντομο σχόλιο. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω ότι είναι ενδιαφέρον και σημαντικό να υπάρχει αυτό το παρατηρητήριο αγοράς ε, ηχθειακών ε, προϊόντων. Το θέμα είναι τι στόχο έχει αυτό το παρατηρητήριο. Πρέπει να ορίσουμε καλύτερα μια πραγματικότητα η οποία σε γενικές γραμμές είναι γνωστή και όλα αυτά τα θέματα τα γνωρίζουμε εδώ και αρκετό καιρό. Αυτά δηλαδή που θέλει να παρατηρήσει το παρατηρητήριο. Είναι απαραίτητο λοιπόν να υπάρχει παρέμβαση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτροπής. Ένα παρατηρητήριο βεβαίως εξορισμού ε, παρατηρεί καταστάσεις και μας ε, επιτρέπει να ε, γνωρίσουμε την πραγματικότητα με τρόπο περισσότερο ακριβή. Είναι λοιπόν σημαντικό να παρέμβει κανείς ε, σε μια τέτοια πραγματικότητα γιατί η κατάσταση είναι δραματική, υπάρχει κρίση στον τομέα, οι τιμές ε, των προϊόντων είναι πολύ χαμηλές. Ε, μιλάμε λοιπόν για μια γνωστή τάση που είναι όμως σημαντικό να παρέμβουμε. Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο σχόλιο που ήθελα να κάνω, είναι ότι ε, πρέπει να παρέμβουμε. Και τώρα θα ήθελα να κάνω κάποιες ε, ερωτήσεις ε, μετά την ομιλία σας. Ομολογώ ότι είχα κάποια δυσκολία να κατανοήσω τις πληροφορίες που μας δώσατε. Υπάρχουν διάφορα επίπεδα στα οποία καλείται να παρέμβει το παρατηρητήριο. Παραδείγματο χάρη ε, σε επίπεδο ανάλυση, ε, δηλαδή σε επίπεδο εβδομαδιαία ενημέρωση για τα προϊόντα. Αυτό είναι το πρώτο επίπεδο. Ε, ένα δεύτερο επίπεδο είναι μηνιαίε πληροφορίες σχετικά με τι τάσει της αγοράς και στο τρίτο επίπεδο εκεί γίνεται λόγος ε, για περισσότερο ε, διαρθρωμένα στοιχεία τα οποία όμως ε, απορρέουν από κατώτερα επίπεδα ενημέρωσης. Έχουμε διαρθρωτική ενημέρωση η οποία απορρέει από την ενσωμάτωση βασικών χαρακτηριστικών και δεδομένων για την αγορά. Διερωτώμε λοιπόν Πώς μπορούμε να έχουμε καλή κάλυψη ε, δομικών ή διαρθρωτικών ε, στοιχείων να γνωρίζουμε τις ε, τάσεις της αγοράς. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι πολλές φορές τα στοιχεία είναι ελλειπή και διερωτώμε πώς είναι δυνατόν να έχουμε καλύτερα στοιχεία γιατί επαναλαμβάνω πολλές φορές ε, τα στοιχεία είναι ελλειπή. Ξέρω αν γίνομαι κατανοητός. Και ίσως μπορείτε να μας δώσετε και κάποιες ε, συγκεκριμένες ε, διευκρινήσεις. Όσον αφορά τώρα τις πηγές ενημέρωσης, θα ήθελα να κατανοήσω καλύτερα ποιοι είναι οι ιδιώτες ε, από τους οποίους αποκτάτε τις πληροφορίες. Ίσως να μην θέλετε να τους αποκαλύψετε, αλλά καταλαβαίνετε ότι θέλουμε να γνωρίζουμε ποια είναι τα μέσα με βάση τα οποία αποκτά κανείς τις πληροφορίες. Τι είδους πληροφορίες μπορεί κανείς να ε, περιμένει, κυρίως ε, τα μέσα, με ποια μέσα αποκτώνται οι πληροφορίες. Και κατόπιν μια άλλη ερώτηση που αφορά στο χρονοδιάγραμμα. Αν κατάλαβα λοιπόν καλά, τέλος του 2011 και αρχές του 2012 θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα του παρατηρητηρίου με πληροφορίες ε, οι οποίες ε, θα τεθούν στη διάθεσή μας. Και μας είπατε ότι το 2012 ε, θα περάσετε σε μία πειραματική φάση. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, πότε θα μπορούμε να έχουμε πληροφορίες εκ μέρους του παρατηρητηρίου. Σας ευχαριστώ. Η ε, κυρία Μπαρέ. Εάν επιβιώσουμε από το πολύ μεγάλο ψύχος που έχει μέσα στην αίθουσα. Ναι, το υποφέρουμε από χθε αυτό το κρύο εδώ μέσα. Λοιπόν, είναι σημαντικό το παρατηρητήριο. Εσείς βάλατε ένα ερωτηματικό βέβαια στα επικυρωμένα δεδομένα. Εμένα με ανησυχεί το θέμα των δεδομένων. Με ανησυχεί η ομοιογενοποίηση των κριτηρίων, ο τρόπος επιλογής, η συλλογή δεδομένων και η επεξεργασία τους. Κάθε χώρα θα ακολουθήσει ένα διαφορετικό τρόπο. Πώς θα ελέγξουμε ότι είναι ομογενοποιημένα τα στοιχεία. Το παρατηρητήριο παρατηρεί, το λέει και το όνομά αλλά ε, επίσης θα γνωμοδοτεί. Δεν ξέρω κατά να αυτά τα... Ε, μάλλον θα ε, βοηθά στο σχηματισμό απόψεων. Πώς ε, θα αποφύγουμε το να χρησιμοποιηθεί για την παραπλάνηση και δεν θα χειραγωγηθεί. Πώς μπορούμε να το αποφύγουμε. Είναι εύκολο. Πάρα πολύ εύκολο να χειραγωγηθούν τα στοιχεία. Και αυτοί πάροχοι δεδομένων που θα τα πουλάνε, γιατί το ξέρουμε, υπάρχουν τέτοιοι σε διάφορες χώρες. Και ξέρουμε και τι τάσεις έχουν, είναι μεροληπτικές. Και γι' αυτό δημιουργούν, σχηματίζουν, μορφώνουν απόψεις, γνώμες. Νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε και να αποκτήσουμε μια μεγαλύτερη γνώση για το θέμα και να μας δώσετε και κάποιες λεπτομέρειες, κάποιες απεξηγήσεις για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Δεν βλέπω ότι ε, δεν βλέπουμε να υπάρχει κάποιο άλλο λιπρόδο. Θα ήθελα και εγώ να προσθέσω κάποια ερωτήματα για τα δεδομένα. Ρώτησαν και άλλοι, δεν θα επεκταθώ. Σε ό,τι αφορά όμω τα αυτά τα προϊόντα που λέτε, που θα μας δίνετε σε εβδομαδία βάση, τι τιμέ κτλ. Μιλήστε για τα πιο αντιπροσωπευτικά προϊόντα. Για πόσα περίπου μιλάμε. Τι κριτήρια θα χρησιμοποιήσετε για την επιλογή αυτών των προϊόντων. Δεν ξέρω, μιλάμε για 50.000 ή για 2 ας πούμε. Ε, δεν αναφέρεται περίπου για ποια ποσότητα, για ποιο αριθμό μιλάμε. Επίσης, έχετε επιλέξει για την πρώτη φάση πέντε αγορές, πέντε βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο. Γιατί, εντάξει, καταλαβαίνω ότι και για μένα κάποιες είναι σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές, για κάποιες άλλες ε, έχω κάποιες αμφιβολίε. Αλλά σε ποια κριτήρια βασιστήκατε για να επιλέξετε τις πέντε αυτές αγορές, τις πέντε αυτές χώρες. Δεν έχω άλλες ερωτήσεις. Κύριε Ραμπό, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Μάλλον εγώ δεν τα είπα καλά. Έχουμε στοχεύσει πέντε κράτη-μέλη. Είπα ότι είναι πραγματικότητα τέτοια. Έχουμε κάποιες συγκεκριμένες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες αυτή τη στιγμή μόνο σε πέντε χώρες. Για το χονδρικό εμπόριο συγκεκριμένα τρία κράτη-μέλη είχαν ε, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία. Χονδρικό εμπόριο, στοιχεία δηλαδή. Ένα συγκρίσιμο σύστημα, όχι όμως ταυτόσιμο, έχει το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό ήθελα να πω. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να απαντήσω συνολικά στα διάφορα ερωτήματα. Πρώτον, σε ό,τι αφορά τον όγκο, τον αριθμό των πληροφοριών. Σε συνάρτηση με τα μέσα, δηλαδή αν θέλουμε ένα μέσο εβδομαδιαίας ενημέρωση όπως σας είπα, που θα προορίζεται κυρίως ε, για τον κλάδο, για τους αγοραστές, ώστε να έχουν μια ιδέα για τις τάσεις. Αν επιλέξουμε αυτό, τότε θα επεξεργαστούμε κάποια προϊόντα αναφοράς. Λοιπόν, ποια είναι η μέθοδος. Θα δούμε ποια είναι τα προϊόντα αναφοράς που χρησιμοποιούνται επί του στα κράτη-μέλη. Δεν θα υπάρχει αρχικά μία πλήρης αρμονία σιγά-σιγά. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι πάντοτε να έχουμε το ίδιο προϊόν και να το παρακολουθούμε σε εβδομαδιαία βάση σε όλη τη διάρκεια του έτους και επί σειρά ετών. Αυτή είναι η ιδέα μας, να υπάρχει μια συνέχεια στην παρατήρηση. Και φυσικά δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να καλύψουμε διεξοδικά, εξαντλητικά όλα τα προϊόντα. Τα βασικά προϊόντα θα καλύψουμε. Δεύτερο επίπεδο τώρα. Μηνιαίες αναλύσεις. Εκεί, αντιθέτω, στόχο μα είναι να είμαστε όσο δυνατόν πιο διεξοδικοί και πλήρει γίνεται. Γιατί θέλουμε να έχουμε ανάλυση των μηνιών πληροφοριών για να έχουμε μια σαφή εικόνα τη εξέλιξη, του πώ εξελίσσεται η αγορά ή οι αγορέ των, ε, ε, των προϊόντων αλληλεία και θετοκαλλιέργεια. Πιο εναρμονισμένη λοιπόν και ευρύτερη γκάμα των πληροφοριών σε σχέση με τα εβδομαδιαία στοιχεία. Ένα άλλο ερώτημα. Πώς θα εργαστούμε. Είπα, εθελοντικά. Εθελοντική θα είναι η βάση. Σίγουρα στην αρχή θα αντιμετωπίσουμε κάποιες δυσκολίες. Δηλαδή να εξηγήσουμε και να γίνει κατανοητό γιατί έχουμε εδώ αυτό το προϊόν, γιατί έχουμε εκεί το άλλο κτλ. Αλλά η συνέχεια είναι το θέμα. Αυτή ε, η συνέχεια θα ε, δώσει και την όλη χρησιμότητα του παρατηρητηρίου. Θα δούμε πώς θα εξελίχνουν τα πράγματα, αλλά επειδή δεν θέλουμε να επιβάλλουμε νέο διοικητικό άχθος, να δημιουργήσουμε νέες υποχρεώσεις ή νέο κόστος, νέες δαπάνες, στις εθνικές δαπάνες, ή τις περιφερειακές δαπάνες, τις τοπικές δαπάνες, θα βασιστούμε στα υφιστάμενα, στα υπάρχοντα. Τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή στη θέση μας νομίζουμε ότι είναι αρκετά για να έχουμε κάτι που δεν είχαμε ποτέ μέχρι τώρα, δηλαδή οικονομική ευφυΐα, για να καταλάβουμε, και νομίζω ότι έτσι απαντώ και σε ένα από τα πρώτα ερωτήματα, για να καταλάβουμε ε, πραγματικά αν υπάρχει κρίση ή όχι. Και αναλυτικά, αλλά και εκ των προτέρων, να έχουμε κάποια στοιχεία ώστε οι λήπτες, αυτοί που λαμβάνουν τις πολιτικέ αποφάσεις, να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα. Δεν θα εργαστούμε μέσα σε καθεστώς ανασφάλειας και αβεβαιότητας, αν λειτουργεί στο παρατήριο όπως λέω. Ούτε με βάση εκτιμήσεις, εντυπώσεις, ούτε θα είναι περιοριστική η άποψή μας. Είναι μια πρόκληση αλλά μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση. Και μαζί και με άλλες συνιστώσεις της κοινή αλληλευτικής πολιτικής νομίζω ότι θα έχουμε μια γενική οικονομική εικόνα της όλης πολιτικής και θα μπορούμε έτσι να λάβουμε τις καλύτερες ε, δυνατές αποφάσεις. Σε σχέση τώρα με τη φύση των πληροφοριών θα δουλέψουμε αναστρώματα πληροφορίες εβδομαδίε για κάποια προϊόντα, ε, μηνιαίες πληροφορίες για κάποια άλλα προϊόντα και πληροφορίες αιτήσεις για κάποια άλλα προϊόντα. Ή ειδικέ αναλύσεις για το σχηματισμό των τιμών. Αυτό θα μπορέσουμε να το κάνουμε, γιατί στόχος μας είναι όλες αυτές τις πληροφορίες να μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε κατά τρόπο ώστε να δώσουμε το ε, ζητούμενο προϊόν. σε ό,τι αφορά τι επόμενε φάσει, μάλλον δεν ήμουν ξεκάθαρο. Δεύτερη φάση είναι η οικοδόμηση του συστήματο. Και η φάση των δοκιμών, ουσιαστικά μιλάμε για μία ε, δοκιμή, γενική δοκιμή, όπου ε, και ο Σύμβουλο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ε, δουλέψουν πάνω σε συγκεκριμένα προϊόντα, με βάση του όρου που σα εξήγησα, για κάποιου μήνε. Για να δούμε αν αυτό λειτουργεί ή όχι. Και εάν δεν λειτουργεί, να κάνουμε τις απαραίτητες προσαρμογές, διορθώσεις, είτε στα εργαλεία αν ένα ζήτημα τεχνικό, πληροφορικής, αν όμως πρόκειται για τη βελτίωση ή τη συνεργασία Κομισιών Εθνικών Υπηρεσιών, θα επικεντρωθούμε σε αυτόν τον άξονα. Η φάση της δοκιμής λοιπόν είναι, έχει ως στόχο στο τέλος να έχουμε κάτι το οποίο πραγματικά θα λειτουργεί, να αρκεί δηλαδή να πατήσεις το κουμπί. Τι θα πει πατάω το κουμπί. Πρώτον, να υπάρχει νομική βάση η οποία θα θεσπίζει την αναγκαιότητα να υπάρχει αυτό το μέσο οικονομικής ευφύειας και νομίζω ή μάλλον ξέρουμε όλοι ότι σε κάποιες εβδομάδες θα διατυπώσει πρόταση μεταρρύθμισης της κοινή ελευθερικής πολιτικής κομισιόν. Και σε αυτό το πακέτο θα υπάρχουν οι διατάξεις οι οποίες θα ε, θεσπίζουν τουλάχιστον την νομιμότητα, ε, αν μη και την πραγματική νομική βάση για αυτό το εργαλείο. Άρα, από το Σεπτέμβριο και μετά θα εργαζόμαστε εκ παραλίλου επί δύο θεμάτων. Πρώτον, τεχνικό, όλος ο τεχνικός φάκελος. ΚΟΖΕΑ και υπηρεσίε της Κομισιόν, φάσεις 2 και 3, και εκ παραλίλου οι συνομοθέτες θα επεξεργαστούν πλέον την δημιουργία αυτού του παρατηρητηρίου ή την αναγκαιότητα να υπάρχει αυτή, ε, αυτό το μέσο οικονομικής ε, στην υπηρεσία των πολιτικών, της πολιτικής. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ρεμπό. Θεωρούμε ότι έχει ολοκληρωθεί το σημείο αυτό. περάσουμε στα διάφορα λοιπόν. Αν δεν υπάρχει κάτι να περάσουμε στο σημείο 14 που είναι οι ανακοινώσεις της Προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις που έλαβαν οι συντονιστές. Έχετε λάβει ε, τις αποφάσεις που λάβαμε χθε. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις μπορούμε να τις θεωρήσουμε εγκεκριμένες. Άρα το μόνο που από μένα να κάνω είναι... Α, συγγνώμη, έχουμε το θέμα του κυρίου Μιλάνα. Το ξέφυγα. Ναι, ε, είναι από το κρύο που κάνει εδώ. Το μόνο που θέλω είναι να φύγω από αυτή την αίθουσα. Έχω ξεπαγιάσει. Λοιπόν, έχουμε πράγματι το θέμα του κυρίου Μιλάνα. Δεν ξέρω ποιος είναι εδώ από την Κομισιόν. Κύριε Μιλάνα, θα σας δώσω εσάς το λόγο καταρχάς και μετά στην Κομισιόν. Επειδή κάνει κρύο θα είμαι και εγώ πολύ σύντομος. Κοιτάξτε, εγώ ασχολούμαι με το θέμα αυτό από το Δεκέμβρη που μας πέρασε και ξεκινήσαμε από μία συζήτηση που έγινε ε, στην Επιτροπή Αναφορών. Είχαμε μία αναφορά ενός πολίτη ο οποίος ρώταγε, ζητούσε να μάθει το λόγο γιατί ε, στα κονσερβοποιημένα ψάρια δεν αναφέρεται η χώρα προέλευσης. Ε, Υπήρχαν δύο γνωμοδοτήσεις από αυτού. Η μία από την, μία πρωτοβουλία από την κυρία Δαμανάκη για το θέμα αυτό ε, και στην πρώτη ερώτηση που ετέθη, η κυρία Νταμανάκη είχε πει ότι θα ασχοληθούμε το θέμα αυτό στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της κοινή ελληνικής πολιτικής, αλλά και στο πλαίσιο άλλων κανονισμών που και αυτοί ε, πρόκειται σύντομα να εκδοθούν. Αυτή ήταν η πρώτη απάντηση που εδώ Δεν ήταν βέβαια ιδιαίτερα ικανοποιητική, παρότι έγινε λόγος για μεταρρύθμιση της ε, κοινή ε, ελληνικής πολιτικής. Εν τω μεταξύ προέκυψε το ατύχημα στην Ιαπωνία και υπήρχε μια δεύτερη δεύτερη ερώτηση. Ε, στην, κατά την ερώτηση αυτή δεν υπήρχε βέβαια η βεβαιότητα ότι τα ψάρια που λέγονται στην Ιαπωνία θα μπορούσαν να καταλήγουν σε κονσέρβες. Όμως, ε, όπως ακούσαμε και σήμερα το πρωί, ε, πέρα από κάποιες απαγορεύσεις είναι δυνατόν να υπάρχει παράνομη αλεία η οποία θα αλλιεύει ψάρια, τα οποία ε, ενδεχομένως να μην μπαίνει σε κονσέρβες ε, στην Ιαπωνία, αλλά σε άλλα μέρη όπως πρέπει τους χάνει στην Παππούα Νέα Και με τον τρόπο αυτό οι συμφωνίες συνεργασίες που έχουμε με την Παππούα Νέα επιτρέπουν στη χώρα αυτή να κονσερβοποιεί ψάρια χωρίς όμως να υπάρχουν εγγύησεις. Άρα δηλαδή τα ψάρια, οι κονσέρβες από εκεί μπορούν να φτάσουν στις διεθνείς αγορές ε, στο σημείο λοιπόν αυτό ρώτησα και εγώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά πόσον έχουν ε, ληφθεί έχει ληφθεί μέρημνα εγγυήσει για τέτοιου είδου ε, προϊόντα. Σήμερα βέβαια το θέμα είναι θέμα ασφάλεια, αλλά τίθεται και το θέμα χρήση, ε, τίθεται και θέμα έλλειψη νομοθετική που δεν προβλέπει την ένδειξη προέλευσης του προϊόντος που βρίσκεται μέσα σε κονσέρβα του, τόνου συγκεκριμένα. Δεν λέει από πού προέρχεται το ψάρι, λέει που έγινε η κονσερβοποίηση. Με τον τρόπο λοιπόν αυτό μπορούν να προκύψουν καταστάσεις ε, που σίγουρα δεν είναι σωστές. Η Ευρωπαϊκή λοιπόν Επιτροπή απάντησε ότι στην Ιαπωνία ε, είναι τα πάντα υπό έλεγχο, τα ακούσαμε αυτό και σήμερα το πρωί, και απάντησε ε, ο Επίτροπος Νταλή ότι όσον αφορά το θέμα αυτό, μάλλον ομολόγησε ότι δεν γίνεται αναφορά του προϊόντος το οποίο βρίσκεται μέσα στην κονσέρβα. Εγώ ήθελα να θίξω το θέμα αυτό και ευχαριστώ τη Γραμματεία και τον Πρόεδρο που με επέτρεψαν να το θίξω το θέμα, γιατί κατ' εμέ ε, αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Υπάρχει θέμα υγιεινής, ε, υγείας ε, γενικότερα. Ακούσαμε βέβαια σήμερα το πρωί ότι αυτό αντιμετωπίζεται με το ότι μπλοκάρεται η αλία σε αυτές τις περιοχές. Υπάρχει βέβαια η παράνομη αλία. Υπάρχει και ένα δεύτερο θέμα, ότι τελικά στις αγορές φτάνουν προϊόντα αλίας τα οποία έχουν συσκευαστεί σε χώρο προέλευσης που δεν έχει σχέση με την αλία αλλά με τη μεταποίηση. Και τρίτον, η συμφωνία με την ε, Παππούα Νέα Γουινέα, η συμφωνία αυτή είναι εκείνη που ε, προσφέρει ιδιαίτερε δυνατότητε στη χώρα αυτή για να μπορούν τα προϊόντα της χώρας να φτάνουν στις δυτικέ αγορές. Ήθελα λοιπόν να θίξω το θέμα αυτό για να ακούσω την άποψη της Επιτροπής και ενδεχομένως και για να δούμε τι θα κάνουμε. Γιατί παρεξία έγινε και στην Επιτροπή Αναφορών και η Επιτροπή Αναφορών δεν το έκλεισε το θέμα, το άφησε ανοιχτό τόσο όσον αφορά σε θέματα που έχουν σχέση με την ενημέρωση των καταναλωτών, όσο και όσον αφορά σε θέματα που αφορούν στην διατροφική ασφάλεια. Ο κύριος Φλούε από τη ΓΑΜΑ ΣΑΚΟ είναι εδώ. Έχετε το λόγο εκ μέρους της Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ασχολούμαι με θέματα ασφάλειας των τροφίμων και η ερώτηση αφορά την υπηρεσία μου. Έχοντας ακούσει λοιπόν το όλο ιστορικό, φοβάμαι ότι το μόνο που μπορώ να σας πω, ε, αυτό μπορώ να πω έχει σχέση με το πυρηνικό ατύχημα στη Φουκοσίμα. Είναι αλήθεια ότι σας απαντήσαμε καθυστερημένα και γι' αυτό υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Κυρίως το ότι η Ιαπωνία είχε ε, να λάβει πάρα πολλά μέτρα το, από το Μάρτιο μέχρι το Μάιο ε, για θέματα ασφάλειας ε, τροφίμων σε σχέση με την Ιαπωνία. Πάνω από 20 κοινοβουλευτικές ερωτήσεις τέτοισαν σε σύντομο χρονικό διάστημα που είχαν σχέση με το ενδεχόμενο ραδιενέργειας σε τρόφιμα στην Ιαπωνία λόγω του πυρηνικού ατυχήματος. Βεβαίως σημαντικό είναι ότι τα μέτρα ελήφθησαν έγκαιρα μετά ε, το πυρηνικό ατύχημα στη Φουκοσίμα στις 11 Μαρτίου. Ήδη στις 15 Μαρτίου η Επιτροπή συνέστησε ε, στα κράτη-μέλη μέσα από το σύστημα ταχείας ε, προειδοποίησης, ενημέρωσε λοιπόν τα κράτη να κάνουν τους απαραίτητους ελέγχους για την ανείχνευση ραδιενέργειας στα τρόφιμα. Ε, αργότερα, πάλι το Μάρτιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τον κανονισμό 297 του 2011, όπου προβλέπονται ιδιαίτερες ε, προϋποθέσεις για την εισαγωγή τροφίμων από την Ιαπωνία. Ο κανονισμός αυτός ε, έχει ήδη τροποποιηθεί δύο φορές για να μπορεί να λάβει υπόψη του τις εξελίξεις, δηλαδή στις 11 Απριλίου και στις 31 Μαΐου. Στις 16 Απριλίου του 2011, ε, πέρα από τα μέτρα που ελήφθησαν και μετά από πληροφορίες ε, για διαρροή ε, πυρηνικής ραδιενέργειας στον Ατλαντικό, η Επιτροπή συνέχισε στα κράτη-μέλη να ελέγχουν τον εντοπισμό ιωδίου και σίου των ενδεχόμενων υπαρξευτών των ε, προϊόντων ε, σε ε, αλληλευτικά προϊόντα κυρίως από τις ζώνες 61, 67, 71 και 77 και αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην αλληλευτική ζώνη 61. Αυτό λοιπόν συζητήθηκε εκτενώς με εκπροσώπους των κρατών μελών στην μόνιμη επιτροπή για την ασφάλεια τροφίμων. Αυτή λοιπόν η σύσταση συμπληρώθηκε από αξιολόγηση κινδύνου για το ενδεχόμενο μόλυνσης από ε, ραδιενέργεια στα προϊόντα λίας στον Ειρηνικό. Και ακολούθησε και ε, δεύτερη σύσταση για τον ε, έλεγχο και έλεγχο ραδιενέργειας σε προϊόντα όπως είναι η το σκουμπρί, οι ε, σαρδέλες και πολλά άλλα προϊόντα. Είχαμε λοιπόν πάρα πολλούς ε, ελέγχους για τον εντοπισμό ε, ραδιενέργειας σε ψάρια από τον Ατλαντικό και όλα τα δείγματα κατέδειξαν ότι δεν περιλάμβαναν ραδιενέργεια, μόνο σε λίγα δείγματα εντοπίστηκαν πολύ χαμηλά επίπεδα ραδιενέργειας, πολύ κοντά στο ανώτατο επιτρεπτό όριο. Για να ολοκληρώσω λοιπόν, αναγνωρίζουμε ότι σας απαντήσαμε καθυστερημένα αλλά ελπίζω να κατανοείτε ότι αυτό οφείλεται ε, στο ότι οι υπηρεσίες ε, είχαν ε, πολλή δουλειά εκείνη τη συγκεκριμένη περίοδο και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι λήφθησαν τα απαραίτητα μέτρα. Επειδή λοιπόν ε, δεν είμαι εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης ε, για την θάλασσα γενικότερα, λυπάμαι που δεν μπορώ να απαντήσω σε άλλες πτυχές της ερώτησής σας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σαραμπό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σε πληρωματικά, να πω καταρχάς ότι επιβεβαιώνω και εγώ ότι είχαμε πολύ καλή συνεργασία με τη ΓΑΜΑ Σάνκο και άλλες υπηρεσίες και θέλω να υπογραμμίσω το εξής. Σε συμπλήρωμα όσων υπάρχουν σε ό,τι αφορά την υγειονομική προστασία υπάρχει ένα μέσο ελέγχου των εισαγωγών. Πιστοποίηση IUU, το ξέρετε όλοι. Σε συνεργασία με τους συναδέλφους από τη ΓΑΜΑΔΕΛΤΑ ΣΑΝΚΟ και τη ΓΑΜΑΔΕΛΤΑ ΤΑΞΟΥΝΤ ακριβώς τη στιγμή που εστέλλονταν ε, και οι κοινοποιήσεις αυτές χρησιμοποίησαμε αυτό το κύκλωμα έγκαιρης προειδοποίησης αλλά και το ΣΥΡΚΑ για να ενημερώσουμε τους τελωνιακούς. Είπαμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα έγγραφο το οποίο συνοδεύει όλα τα αλληλευτικά προϊόντα. Λέγεται πιστοποιητικό IUU και σε αυτό υπάρχουν βασικά στοιχεία τα οποία μπορούν να λύσουν τα προβλήματα που ανέφερε ο κύριος Μιλάν. Όχι το προϊόν, την προέλευση του ε, προϊόντος ε, που έχει να κάνει με το πλοίο και όχι το μέρος που έχει αλλιευθεί. Αλλά ζώνη αλλιεύσης, ζώνη ΦΑΟ και ημερομηνία αλλιεύσης. Αυτά τα δύο στοιχεία. Άρα όλα τα αλλιεύματα που μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνοδεύονται από αυτό το έγγραφο. Σε αυτό το έγγραφο λοιπόν υπάρχουν θέσει δύο πληροφορίες. Ζώνη αλλιεύσης και ημερομηνία αλλιεύσης. Εντάξει, συμφωνούμε. Αυτά είναι πολύ σημαντικά στοιχεία. Και όπως έχει αναφέρει και η κυρία Δαμανάκη, στην Επιτροπή σας νομίζω, είχε λάβει την πρωτοβουλία να υπενθυμίζει στους τελωνιακούς υπαλλήλου ε, των υπηρεσιών υγείας ότι υπάρχει αυτό το μέσο που μπορεί να διευκολύνει και τις δικές τους έρευνες για την προέλευση και το, την καταγωγή αν θέλετε, το origin και ε, την, την προέλευση πάνω των προϊόντων. Με τις ε, χώρες της περιοχής που αναφέρατε θα ε, υπογράψουμε ε, τις ρυθμίσεις αλλά αυτό δεν τις ε, απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις που έχουν αλλά μπορούν να διεισδύσουν αν θέλετε και να πουλήσουν τα προϊόντα τους στις αγορές υποχρεωτικά όμως πρέπει να τηρούν τις δεσμεύσεις υγιεινής Υπάρχουν κάποιες δασμολογικές ε, διευκολύνσεις, αλλά καμία παραχώρηση δεν γίνεται σε ό,τι αφορά το σεβασμό των υγειονομικών κανόνων ή των κανόνων που επιβάλλονται από την κοινοτική νομοθεσία σε σχέση με την πιστοποίηση και δι' την πιστοποίηση για την παράνομη λαθρέα δηλαδή αλία. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα αυτά που μας είπατε, αλλά όλα αυτά μας είπατε τα ξέραμε κατά λέξη. Δηλαδή, το πρόβλημα εξακολουθεί να είναι το εξής, ότι αν υπάρχει τόνος που αλλιεύεται και μπαίνει στην κονσέρβα στην ε, Νέα Γουινέα Παπουασία, η κονσέρβα αυτή μπορεί να φτάσει στις αγορές μας χωρίς να ξέρουμε από πού προέρχεται, ότι πρόκειται από ένα συγκεκριμένο σημείο ζώνη αλίας. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά το Ιαπωνικό ατύχημα σωστά συμπεριφέρθηκε. Πολύ σωστά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έφτιαξε ένα δίχτυ προστασίας. Όμως η ίδια η Επίτροπος, η κυρία Ανταμανάκη, πριν από δύο μήνες μου είπε ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα χωρίς να υπάρχει ένδειξη προέλευσης να φτάσει ένα προϊόν στις ε, αγορές μας. Γιατί σας λέω η ένδειξη αφορά τον συσκευαστή και όχι το προϊόν το οποίο είναι μέσα στο κουτί, στην κονσέρβα. Ε, και μην ξεχνάμε όμως ότι αυτό είναι το θέμα, ότι το προϊόν μέσα στην κονσέρβα μπορεί να είναι μολυσμένο. Εμείς λοιπόν οι καταναλωτές της Ευρώπης, ε, εμείς το Ευρωπαϊκό Οικονομικό Σύστημα δεν μπορούμε να ξέρουμε από πού προέρχεται το προϊόν ε, που βρίσκεται μέσα στην κονσέρβα. Άρα δηλαδή φτάνουμε στο εξή. Οφείλουμε να πούμε και στην Παππούα Νέα Γουινέα ότι Ξέρετε σήμερα τόνος που αλλιεύεται στις Ηνωμένε Πολιτείες μπορεί να μπει σε κονσέρβα. Έχουν γίνει πάρα πολλές παρεμβάσεις από την πρόεδρό μας επί του θέματος αυτού από τι ε, Ηνωμένε Πολιτείε. Πάει στην Παππούα Νέα και μετά ε, φτάνει στι Ηνωμένε Πολιτείε. Και τι ξέρουμε εμεί, ξέρουμε ότι έρχεται από την Παππούα Νέα. Όχι όμω από τι Ηνωμένε Πολιτείε, αυτός λοιπόν ο κύκλος ζωής ε, αφορά προϊόντα που μπορούν να έρχονται από πουδήποτε. Άρα δηλαδή ε, γιατί να μην έρχονται και από παράνομη αλία ε, στην περιοχή της Πουκοσίμα. Θα ήθελα να προσθέσω το εξής. Νομίζω υπάρχει ένα ζήτημα... Α, η κυρία θέλει το λόγο. Ε, thank Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα και πολύ πολύπλοκο. Διότι υπάρχουν πολλές ε, γάμα δέλτα που εμπλέκονται και πολλά νομοθετήματα. Εγώ θα ήθελα συγκεκριμένα να εστιάσω ε, στη γάμα δέλτα Μάρη που μας είπε εκπροσωπός της ότι πράγματι υπάρχει η αναφορά της γεωγραφικής ζώνης σε όλα τα προϊόντα τα οποία εισέρχονται στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπατε ζώνη ε, του ΦΑΟ και των ε, παγκόσμιων ε, υδάτων ωκεανών. Τι είναι υποχρεωτικό να αναφέρεται για τον βορειο ανατολικο Ατλαντικό, ΦΑΟ δηλαδή. 13 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα. Αυτή είναι η έκταση της ζώνης από την Βόρεια Νορβηγία μέχρι το Βυσκαϊκό κόλπο και στον Ατλαντικό, στη Μέση του Ατλαντικού. Δεν είναι τόσο ξεκάθαρο και συμφωνώ από κάθε πλευρά για την ανείχνευση παράνομης αλίας, ήταν και από των καταναλωτών και ούτω καθεξής, πρέπει να αναγράφονται πολύ περισσότερες λεπτομέρειες για τη γεωγραφική περιοχή και όχι μόνο ε, η ζώνη ΦΑΟ. Αυτό είναι το σχόλιο μου και νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε και στην κοινή οργάνωση αγοράς και στο πλαίσιο της μεταρρυθμίσης της κοινής αλληλευτικής πολιτικής. Πρόεδρος, πράγματι υπάρχει ένα πρόβλημα που είναι η επισήμανση, η ετικετοθεσία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μια μελέτη και μια από τις που εγώ διάβασα είναι ακριβώ αυτή με τις ε, διαβόητες ζώνες ε, ΦΑΟ. Υπάρχουν υπάλληλοι της ΦΑΟ που καταλαβαίνουν δεν καταλαβαίνουν τις ετικέτες ε, αυτές. Λοιπόν, πρέπει να λυθεί αυτό το ζήτημα και πρέπει να το δούμε στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της κοινή οργάνωσης αγοράς. Είναι ένα από τα σημεία κλειδιά του όλου πακέτου της μεταρρύθμισης που πρέπει να το λύσουμε εδώ. Όλες λοιπόν τις αδυναμίες και τις ελλείψεις πρέπει να τις επισημάνουμε. Και μία από τις αδυναμίες είναι αυτές οι ζώνες φάου που δεν τις καταλαβαίνει κανένας. Και έχουμε τώρα το πακέτο της μεταρρύθμισης και το θέμα της ετικετοθεσίας, της για να μην μιλήσω για, την, για το eco-label, ε, που το έχει ξεχάσει πια η Κομισιόν, αυτά πρέπει να τα επισημάνουμε. Το θέμα της ετικετοθεσίας εγώ θέλω να το ξανά επισημάνω. Πρέπει να βελτιωθεί η επισήμανση, αυτό είναι σαφές. Τι ζώνε ΦΑΟ, ε, όλο ο κόσμο τι ε, κατηγορεί κατά κάποιο τρόπο. Είναι προφανέ ότι δεν είναι ξεκάθαρε. Τώρα, το θέμα της υγείας, το υγειονομικό, ναι, υπάρχουν ε, καλοί ή κακοί έλεγχοι, κάποιες φορές αποτυγχάνουν, αλλά υπάρχει ένα σύστημα, υπάρχει το σύστημα ε, μέτρων υγειονομικού ελέγχου. Νομίζω ότι το θεμελιώδες πρόβλημα είναι με τις ετικέτες. Αυτό το πρόβλημα πρέπει να το λύσουμε και πρέπει να το λύσουμε τώρα, γιατί έπεται η μεταρρύθμιση. Εκτός, σχολείου, μικροφώνου το δεν ξέρω, αλλά πρέπει να λυθεί αυτό το θέμα, λέει πρόεδρο, και έχουμε τώρα τη δυνατότητα, γιατί έρχεται μεταρρύθμιση και μπορούμε να το επισημάνουμε. Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο, ίσω να έχει να πει η Κομισιόν. Επαναλαμβάνω, σε μια μελέτη επιπτώσεων που κάνατε στην Κομισιόν αναλύεται ακριβώ αυτό το θέμα με τι ζώνε ΦΑΟ, που δεν έχει κανένα απολύτω νόημα, καμία απολύτω χρησιμότητα. Λοιπόν, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Θέλω να σα ευχαριστήσω όλου, τον κύριο Ρεμπό, τον κύριο Φλούε πήγαμε Σάνκο. Και έτσι περνάμε στο τελευταίο σημείο τη διάταξη. Προσεχή συνεδριάση. Λοιπόν, προσεχή συνεδρίαση στι Βρυξέλλε, 12 και 13 Ιουλίου. Τέλος τη συνεδρίασης. Παγώσαμε.